Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε να ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίασή μας. Θεωρώ ότι η μερίσια διάταξη έχει εγκριθεί. Ωραία, ευχαριστώ. Οπότε προχωρούμε ευθύ αμέσω στο πρώτο μας σημείο, ο οικονομικός διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με τον Πιέρ Καρλο Παντοάν, υπό την ιδιότητά του ε, εξερχομένου Πρόεδρου του ΕΚΟΦΗΝ και Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας. Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τη μετρική μου γλώσσα σήμερα. Εκτάκτος, να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Να ευχαριστήσω την Ιταλική Προεδρία για τη συνεργασία και για το ρόλο που έχει φέρει πέρα ως τώρα με ένα εξάμεινο που ξεκίνησε αμέσως μετά τις ευρωεκλογέ, ένα εξάμεινο που η νομοθετική δραστηριότητα που αναλαμβάνουν οι εξάμενες προεδρίες μετά τη Λισαβόνα ήταν μια πρόκληση πολύ σημαντική. Θεωρώ ότι τα όσα κατάφερε η Ιταλική Προεδρία ήταν ε, άκρο σημαντικά. Μας επέτρεψε να ολοκληρώσουμε πολλά νομοθετικά θέματα και το σχέδιο κάποια ιδιαίτερα εύστοχα και φαντάζομαι ότι ο Υπουργό ε, πάντω αν θα τα αναφέρει. Ε, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ, αλλά είναι σημαντικότατα νομοθετικά θέματα που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την ε, εξέτασή τους μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Στην ουσία δύο μήνες διαπραγματεύσεων. Και εκτιμήσαμε και τον τρόπο με τον οποίο η Ιταλική Προεδρία μας ε, έκανε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία υλοποίησης για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης, που είναι και καρπός της δικής μας ε, διαμεσολάβησης και προσπάθειας. Νομίζω ότι και η δική μας η Επιτροπή έχει δώσει την πολύτιμη συμβολή της σε αυτό το έργο. Θεωρώ σημαντικό ότι η Ιταλική Προεδρία κατάφερε να προβλέψει και θέματα γενικότερου ενδιαφέροντα ε, στην πολιτική οικονομική λίστα προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, όπως το θέμα των επενδύσεων. Το τι σημαίνει να αξιοποιούμε καλύτερα την ευελιξία που προβλέπει το Σύμφωνο σταθερότητα. αύριο θα δούμε και τα δύο αυτά θέματα και η Επιτροπή μα θα εξετάσει τον κανονισμό, την πρόταση κανονισμού για τους κανόνες ευελιξίας Νομίζω ότι εδώ η Ιταλική Προεδρία συνέβαλε τα μάλα στην ε, πρόθεση των θεμάτων αυτών. Όμως τώρα να δώσω τον λόγο στον ε, Υπουργό Πάντουαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια, για τη δουλειά της Ιταλικής Προεδρίας. Θα θεωρήσω ότι είναι και προσωπικές ευχαριστίες, αλλά βεβαίως και προς όλη την ομάδα συνεργατών της Ιταλικής Προεδρίας που εργάστηκαν ελπίζω αποτελεσματικά. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, σα ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να συμμετάσχω στι εργασίε τη Επιτροπής σα. Εκτίμησα ιδιαίτερο την επικοδομητική σχέση που είχαμε του τελευταίου έξι μήνε. Μα επέτρεψε να καταλήξουμε σε σημαντικότατα αποτελέσματα στο πέρας της Ιταλικής Προεδρίας θεωρώ σημαντικό να κάνω μια ανασκόπηση στα αποτελέσματα που πετύχαμε και στα βήματα προόδου που επιτελέστηκαν. Αλλά κυρίως να θυμίσω αυτά που κατά την άποψή μου ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να διατηρήσουμε για το μέλλον. Από τον περασμένο Ιούλιο είχα αναφέρει ποια θα είναι η προσέγγιση της Ιταλικής Προεδρίας για να στηρίξουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Που θα βασιζόταν σε τρεις πυλώνες. Τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις, τις επενδύσεις και μια βαθύτερη ολοκλήρωση των αγορών. Αυτοί οι πυλώνες ενισχύονται ε, αμοιβαίως και θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε μια στρατηγική συνεπή με μεταρρυθμίσεις την αγορά των εμπορευμάτων και υπηρεσιών, την αγορά εργασίας, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, ώστε να δημιουργηθεί ανταγωνιστικότητα και ευνοητόρο κλίμα για τις ευκαιρίες επενδύσεων. Οι επενδύσεις επιτρέπουν να εδρεωθούν τα θετικά αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων, στηρίζουν την ζήτηση μεσοπρόθεσμα και επιτρέπουν να αυξηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης μέσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ε, οι υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές ενισχύουν περαιτέρω την ζήτηση, την ε, ανάπτυξη και την ε, μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου η συνένεση για αυτή τη στρατηγική επιβεβαιώθηκε και βάσει των προσανατολισμών της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το μακροοικονομικό όμως σκηνικό υποβαθμίστηκε περαιτέρω. Επιδεινώθηκε διότι οι κίνδυνοι αποπληθωρισμού και οι χαμηλότερες επιδόσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών ε, έγιναν πραγματικότητα με ποσοστά ανεργίας που παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Η αποτελεσματική μας απάντηση για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις τάσεις ήταν πήγουσας ανάγκης. Υπάρχει λοιπόν λόγος να συνεχίσουμε μια διαρθρωμένη, ένα διαρθρωμένο θεματολόγιο μεταρρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Και αυτό το, ε, σε αυτό συνενούν όλοι. Η συνεργασία των Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωκοινοβούλιο είναι θεμελιώδης σημασία. Οι συζητήσει στο Συμβούλιο έδειξαν την ανάγκη να ενισχύσουμε την ανάληψη ε, ευθύνη από τα κράτη-μέλη αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Διαδικασία μπορεί να παίξει αποφασιστικότερο ρόλο ώστε να επιβεβαιώσουμε την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που υλοποιούνται. Λόγου χάρη, λαμβάνοντα υπόψη πολιετή χρονικού ορίζοντε, απαραίτητου για την πλήρη υλοποίηση και την εκδίπλωση των θετικών αποτελεσμάτων των μεταρρυθμίσεων. Ενθαρρύνοντα εθνικά προγράμματα ευρέω φάσματο, ώστε να καταλήξουμε σε αποτελεσματικότερα βήματα το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι το σωστό πλαίσιο ώστε να δούμε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ χωρών και να ευρεώσουμε τα θετικά αποτελέσματα με προστιθέμενη αξία, συντονισμένε προσπάθειες και ταυτόχρονες, ώστε να ενισχύσουμε τους δεσμούς και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ χωρών η Ιταλική Προεδρία προχώρησε με την απόφαση να έχουμε ένα θεματολόγιο και μια λίστα προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις με μια δύναμη κρούσης και ε, τις επενδύσεις να αναλαμβάνονται από την ΕΚΤ ώστε τα κράτη-μέλη να εντοπίσουν συγκεκριμένα επενδυτικά προγράμματα και ενδεχόμενους θεσμικούς, οικονομικούς ε, και θεσμικούς φραγμούς που μπορεί να μην επιτρέπουν την εύκολη υλοποίηση. Το αποτέλεσμα των εργασιών της ε, Task Force παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο και είναι ένα σημαντικό σημείο αφετηρίας για να αναπτυχθούν καινοτόμα προγράμματα ε, ε, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, το Συμβούλιο εξέφρασε τη στήριξή του προς το πρόγραμμα των επενδύσεων για την Ευρώπη, όπως είχε παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ θα ασχοληθεί με τη συνεργασία του με το Κοινοβούλιο, ώστε να δημιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Στατικές Επενδύσεις. Είναι θετική η πρόθεση που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ε, θετική εξέταση των εθνικών συνεισφορών προς το Ταμείο προκειμένου να ενθαρρυνθεί η άμεση συμμετοχή των κρατών μελών. Το πρόγραμμα οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση. Η τάση μείωση των επενδύσεων αναχαιτίζεται και προωθούνται στρατηγικές προτεραιότητες προκειμένου να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πέραν από την κινητοποίηση όμω των ε, κρατικών και ιδιωτικών κονδυλίων, προβλέπονται και άλλα σημεία κλειδιά των μεταρρυθμίσεων προκειμένου να υποστηριχθούν οι επενδύσει. Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντο προκειμένου να κινητοποιηθούν οι μεταρρυθμίσει, στόχο έχουν να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα για τα επενδυτικά προγράμματα. Τα, οι επενδύσει γεννώνται από το συνδυασμό δύο παραγόντων τις ευκαιρίες ε, κερδοφορίας και τις ευκαιρίες να τις αξιοποιήσει κανείς. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν ένα σημείο κλειδί για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Αυτό θα είναι το κομβικό σημείο για να πετύχουμε τους στόχους της Ευρώπης του 2020. Υπ' αυτήν την έννοια ε, απαιτούνται ταχύτερες πρόοδοι στην αγορά των υπηρεσιών, την ψηφιακή αγορά και την, τα βιομηχανικά προϊόντα. Υπ' αυτήν την έννοια καλύτερη συνεργασία με μια στρατηγική ανάπτυξη απαιτεί ε, περαιτέρω βήματα για την ε, Τραπεζική Ένωση για να ξεγιανθούν τα χρηματοπιστωτικά συστήματα και τα προϊόντα που θα επιτρέψουν στα τραπεζικά ιδρύματα να προχωρήσουν. Έτσι, τα συμπεράσματα του ΕΚΟΦΗΝ για την ανάπτυξη όπως εγκρίθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο δίνουν χρήσιμους προσανατολισμούς για τις ε, δέουσες παρεμβάσεις. Προκειμένου να υπάρξουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα μακροπρόθεσμα που να επιτρέψουν τη στηρίξη της πραγματικής οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνέπεια των προτάσεων αυτών, η δημοσιονομική ε, χρηστή διαχείριση και η οικονομική, ε, ο οικονομικός σχεδιασμός επιτρέπουν ε, να γίνουν θετικά βήματα εφόσον υπάρξει και απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισίου η φορολογική διαφάνεια, η, απα... η καταπολέμηση της φοροαπάτης και της φοροδιαφυγής είναι σημαντικά στοιχεία. Το 2014 ήταν ένα σημαντικό έτος για το τέλος του τραπεζικού απορρίτου. Τα διεθνή πρότυπα για την αναυτόματα ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοπιστωτικού και οικονομικού χαρακτήρα ενσωματώθηκε στο κοινοτικό δίκαιο πλέον. Το αποτέλεσμα αυτό είναι μια μεταρρύθμιση διαρθρωτικής σημασίας και διεθνούς εμβέλειας που θα επιτρέπει την καλύτερη συμμόρφωση τον ε, και την παρακολούθηση των ε, όσων συνεισφέρουν οι φορολογούμενοι στα εθνικά και ευρωπαϊκά ταμεία. Ως προς την ε, φοραπάτη, την εικονική μετακίνηση των κερδών που ξεκίνησε να προωθείται από τον ΩΣΑ. Είναι στοιχεία που θα στηρίξουν τους διεθνείς φορολογικούς κανόνες. Στην Ιταλική Προεδρία είχαμε μια βαθιά μελέτη των θεμάτων αυτών και κατά πόσον είναι εύστοχα τα αποτελέσματα Ιδίως η συμπερίληψη ρήτρα κατά της επεξήγησης στην ε, οδηγία μητρικές θηγατρικές εταιρείε είναι ένας από τους φιλοδοξότερους στόχους μας για τους επόμενους μήνες με στόχο να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα φαινόμενα του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, της επιζήμιας φορολογικής ανταγωνιστικότητας και των ε, αθέμητων φορολογικών βάσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαφή αυτή την προοπτική ανακοίνωσε την πρόθεσή της να παρουσιάσει σύντομα μια πρόταση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για, τις, ε, για τους φορολογικούς διακανονισμούς. και αυτό βάσει της ε, νομοθετικής βάσης που προτείνει και το Συμβούλιο. Εδώ θα ξεκινήσουμε από τα όσα όρισε και το ΕΚΟΦΗΝ τον Δεκέμβριο με εργασίες για τους φόρους και τις φορολογικές πληροφορίες με τρόπο συντονισμένο και στη διάρκεια του 2015. Δύο λόγια για τα οικονομικά θέματα. Η ΕΚΤ ανέλαβε τα πλήρη καθήκοντα εποπτείας στο Νοέμβριο. Αυτό είναι αποτέλεσμα της κοινή δουλειάς και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και γι' αυτό μπορείτε να είστε υπερήφανοι. Ο μηχανισμός ενιαίας εποπτείας θα στηρίξει την εμπιστοσύνη του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτό είναι ο πρώτος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης. Αυτός ο ενιαίος μηχανισμός όπου θα ενταχθεί και ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανση. Για να γίνει πλήρως λειτουργικός χρειάζονται και οι κανόνες για τους ε, τρόπους συνεισφοράς των τραπεζών στο Ταμείο Διάσωσης. Εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε και για την της πράξης από την οδηγία για την εξηγέση των τραπεζών με ενιαίους κανόνες για τη λειτουργία του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανση. Η συνεργασία αυτή τη Επιτροπή με την Ιταλική Προεδρία ήταν παραδειγματική, προκειμένου να καταλήξουμε σε ισόρροπε λύσει. Δεν μπορώ να σταθώ με λεπτομέρειε σε όλε τι άλλε νομοθετικέ πράξει για τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Απλώ θα πω ποια ήταν τα σημαντικότερα αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα, χάρη και στην επικοδομητική συνεργασία του Ευρωκοινοβουλίου, πετύχαμε συμφωνία στον κανονισμό για τα ε, μακροπρόθεσμα επενδυτικά ταμεία τη Ευρώπη, τα LTIF. Επίσης, ήταν σημαντική πολιτική συμφωνία που πετύχαμε στον τριμερή διάλογο της 17ης Δεκεμβρίου για τον κανονισμό που αφορά τις διατρα... πολυμερείς διατραπεζικές επιτροπές και τις συναλλαγές πληρωμής πληρωμών μέσω πιστοτικών καρτών. Επίσης, συμφωνία υπήρξε για τον κανονισμό κατά της νομιμοποίησης παρανομών προσόδων, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών ε, μέσω του γκάφη. Τέλος, ε, οριστικοποίησαμε τις θέσεις του Συμβουλίου ως προς τον κανονισμό για, την, ε, ε, για τη δημοσιονομική συνεργασία για τις επιχειρηματικές και επαγγελματικές για τους επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς φορείς για τις πληρωμές και για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εδώ έγιναν θετικά βήματα πρόοδου ως προς την διευθυντική μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα, τα, και τους δείκτε συγκριτική αξιολόγηση που χρησιμοποιούμε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ε, κύριε Πρόεδρε, ε, η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία είναι σημαντικά στοιχεία για την εμπιστοσύνη των, ε, για την λειτουργία των οικονομικών φορέων και των επενδυτών. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο θετικό κλίμα στην Ευρώπη ώστε να έχουμε προοπτικέ ευημερία. Δεδομένη τη βαρύτητα τη κατάσταση, η Ευρώπη, όπω υπενήχθηκα, χρειάζεται ένα θετικό σοκ για να γυρίσει σελίδα πιο γρήγορα. Θα πρέπει λοιπόν η δράση μας να είναι αποφασιστική, διαρθρωμένη και συνεπής. Οι επενδύσεις θα πρέπει να υποστηριχθούν ώστε να υπάρξει ένα σημαντικό αντίκτυπο στην ζήτηση στην αγορά και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη μέσω πρόθεσμα. Ε, το θεματολόγιο των προτεραιοτήτων μα πρέπει να είναι φιλόδοξο και να υπάρξει πυγμή και αποφασιστικότητα μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να συμπληρώσει το εύρο των, των οικονομιών τη Ευρωζώνη ε, μαζί με την θετική ανάπτυξη και τι μεταρρυθμίσει που θα επιτρέψουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα. Είναι θεμελιώδου σημασία να υπάρξει ε, στην πράξη παρακολούθηση ε, των αποτελεσμάτων ε, με τα όσα ορίζει, σε συνέπεια με τα όσα ορίζει και το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Έτσι θα βελτιωθεί το δυναμικό ανάπτυξη τη ευρωπαϊκή οικονομίας και θα αξιοποιήσουμε πλήρω την αξιοπιστία του συστήματο κανόνων μα. Θα επιτρέψουμε να είναι αξιόπιστα τα κρατικά δημοσιονομικά και ε, ε, κρατικές οικονομίες, οπότε να υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις, ε, κινητοποίηση και ε, απασχόληση. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους κανόνες ευελιξίας στα πλαίσια της όλης συζήτησης που θα γίνει τις ερχόμενες εβδομάδες για την αναθεώρηση της διακυβέρνησης ε, ενισχυμένη με το δίπτυχο και εξάπτυχο μέτρων όπου ο ρόλος του Κοινοβουλίου και της δικής σας Επιτροπής είναι θεμελιώδου σημασίας. Και πάλι ολοκληρώνοντας να σας ευχαριστήσω για τον επικοδομητικό σας ρόλο του τελευταίου τους και για ε, την παρουσία σας απόψε. Εύχομαι καλή τύχη στη Λετωνική Προεδρία και ε, κάθε επιτυχία στα βήματα που θα επιχειρήσει. Ευχαριστώ κύριε Παντουάν. Ερωτήσεις και απαντήσεις. Πέντε λεπτά για κάθε ερώτηση αλλά και την απάντησή της. Παύλο θα μιλήσω. Κύριε Υπουργέ, κατά πρώτον συγχαρητήρια για τα επιτεύγματα της Προεδρίας σας. Είχα και εγώ προσωπικό στην ευκαιρία να εργαστώ ως εισηγητής επί ενός εκ των θεμάτων που αναφέρατε. Συγκεκριμένα τις διτραπεζικές ε, ε, χρεώσεις, ε, επιπράξεων με επιστορικές κάρτες κλπ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς και την ομάδα διαπραγματεύσης η οποία τα πήγε εξαιρετικά τουλάχιστον. Έχω κάποιε ερωτήσει για την Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, τι γίνεται στην Ελλάδα, ποια είναι η εντύπωσή σα, ποια είναι η αίσθησή σα και ποια είναι η πρόβλεψή σα για το τι θα μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα. Και κάτι για τη χώρα σα. Δεν είμαι βεβαίω ε, αρμόδιο να αξιολογήσω την κατάσταση στη χώρα σα, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι οι μεταρρυθμίσει είναι σημαντικέ όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό. Θα μπορούσατε λοιπόν να μα πείτε πώ εξελίσσονται, πώ πηγαίνουν οι μεταρρυθμίσει στη χώρα σα και τι είδου αποτελέσματα προσδοκάτε. Τέλος, για το σχέδιο Juncker, σήμερα αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας συζήτησε το σχέδιο Juncker. Πιστεύω ότι η εκτίμηση είναι ότι θα πετύχει με την προϋπόθεση ότι θα επιλέξουμε τα σωστά έργα, θα κάνουμε τις σωστές κινήσεις. Πώς θα γίνει όμως αυτό κατά τη γνώμη σας. Πώ θα επιλέξουμε τα σωστά έργα ώστε να επιτύχει το σχέδιο Juncker. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις σας. Οπότε θα προσπαθήσω να τις απαντήσω μία προς μία. Για την Ελλάδα πρώτα απ' όλα. Ποια είναι η πρόβλεψή μου. Είμαι οικονομολόγος, ε, οπότε καταλαβαίνω ότι δεν, πρέπει να, δεν μου επιτρέπεται να κάνω προβλέψεις. Όμως να σας πω ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα στο χρόνο, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Η χώρα υλοποίησε επώδυνες μεταρρυθμίσεις στον δημοσιονομικό τομέα. Δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν όσον αφορά τη δημοσιονομική εξυγίανση. Όλα αυτά βεβαίως εν μέσω ασθενικής οικονομίας και χαμηλού πληθωρισμού στην Ευρώπη, κάτι το οποίο δεν βοηθάει βεβαίως ε, την βιωσιμότητα του χρέους. Στο πλαίσιο αυτό η ελληνική κυβέρνηση με την πολύτιμη βοήθεια των μελών τη Τρόικας σημείωσε πρόοδο. Πιστεύω ότι μπορεί να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος και προσωπικός Έχω την πεποίθηση ότι η νέα κυβέρνηση, η οποία θα προέλθει από τις προσεχείς εκλογές, θα συνεχίσει στον δρόμο, στον ίδιο δρόμο, συνεχίζοντας δηλαδή την προσπάθεια, τις προσπάθειες των προηγουμένων κυβερνήσεων και μάλιστα θα έλεγα του ελληνικού λαού εν το σύνολο του. Και ότι όλα αυτά θα συνεχιστούν όπως είπα περαιτέρω προσπάθειες και σε πλήρη συμφωνία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου αν θέλετε. Είναι και η ευχή μου και σε ό,τι φορά την Ιταλική κυβέρνηση θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε την συνολική αυτή προσπάθεια Ελλάδας και Ευρώπης. Για την Ιταλία τώρα. Θα έλεγα ότι η στρατηγική της κυβέρνησης είναι σχεδόν αποκλειστικά εστιασμένη στην θέσπιση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στην εφαρμογή τους. Ένα από τα σημεία τα οποία ακούγονται συνεχώς τους τελευταίους δεκαμήνες είναι ότι ξέρετε έχουμε πήξει τις ανακοινώσεις, έχουμε υπερβολικά πολλές ανακοινώσεις αλλά το θέμα είναι ότι Έχουμε μπροστά μας πολλές μεταρρυθμίσεις που τις ανακοινώσαμε αλλά δεν τις υλοποιήσαμε. Και αυτό εξηγεί το γεγονό ότι εδώ και τρία χρόνια περιμένουμε την, τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Χάσαμε ευκαιρίες, δυστυχώς, την δημοσιονομική εξυγίανση. Δεν μεταρρυθμίσαμε την οικονομία. Έπρεπε να κάνουμε λοιπόν μεταρρυθμίσεις και δεν τις κάναμε. Τούτου λεχθέντος Σημειώθηκαν και σημαντικά πρακτικά αποτελέσματα. Τα πετύχαμε χάρη στην Ιταλική Βουλή, χάρη σε αυτούς που τις υλοποίησαν. Μεταξύ άλλων έχουμε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, είναι ο νόμος περί εργασίας, έτσι όπως το ονομάζουμε στην Ιταλία, πολύ σημαντικός νόμος, ο οποίος αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται. Σήμερα ήμουν στο Σάλτσμπουργκ και άκουσα ότι η κυβέρνηση υλοποίησε και άλλον έναν ε, νόμο σχετικά με τα επίδοματα ενεργεία. Αλλά έγιναν και άλλε σημαντικέ μεταρρυθμίσει και άλλε θα γίνουν. Πρόκειται για δημοσιονομικέ μεταρρυθμίσει, όπω είπα. Ένα τομέα στον οποίο αλλάζουμε την διακυβέρνηση, βελτιώνουμε την διαφάνεια, εξασφαλίζουμε συμμόρφωση των φορολογουμένων με την κείμενη νομοθεσία. Τέλος για το σχέδιο Juncker, κοιτάξτε αυτό δεν θέλω να ακουστώ απεσιόδοξο, αλλά θα πάρει χρόνο. Και παρέχομαι στην αρχική μου παρατήρηση. Πρέπει όλοι εδώ να συνεργαστούν. Χρειαζόμαστε πολλές προϋποθέσεις, τους πόρους και σωστή διακυβέρνηση. Είμαι πάντως πεπισμένος ότι ο μηχανισμός επιλογής και υλοποίησης που συνοδεύει τον μηχανισμό θα επικυρωθεί σύντομα και όχι μόνο θα δημιουργήσει ευκαιρίες επενδύσεων αλλά θα βελτιώσει και την απόδοση των επενδύσεων και της δημοσίας διοίκησης ανά την Ευρώπη. Όλοι θα βγουν κερδισμένοι από κάτι τέτοιο. Έτσι θα παρασπούν, όπως είπα, περισσότερα κίνητρα για να υλοποιηθούν επωφελεί για όλε τις επενδύσεις. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά ήταν τρει ερωτήσει σα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ επομένω από του σοσιαλιστές Λίζα Φερέρα. Ευχαριστώ και εγώ θα χρησιμοποιήσω τη μετρική μου γλώσσα. Συγχαρητήρια για την δουλειά της Ιταλικής Προεδρίας. Συγχαρητήρια και στους ε, υπευθύνους που είναι σήμερα εδώ. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα των συνεργατών. Νομίζω ότι το έργο σας ήταν πολύ σοβαρό και υπό αντίξωες συνθήκες. Και αυτές οι αντίξωες συνθήκες ε, είχαν να κάνουν όχι μόνο με το ότι ανανεώθηκαν τα θεσμικά όργανα και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, αλλά και με το ότι η συγκυρία ήταν η μακρά αυτή περίοδος ύφεσης και ανεργίας που έκαναν τα πράγματα πάρα πολύ περίπλοκα. Η Ιταλική Προεδρία πέραν του θεματολογίου που αναφέρατε μπόρεσε να δώσει την απαραίτητη έμφαση στις επενδύσεις και στην ανάγκη των επενδύσεων αλλά και στην ε, ανάγκη να εξισορροπηθούν τα κρατικά δημοσιονομικά με τις επενδύσεις. Νομίζω ότι άρχισαν τα πρώτα βήματα προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις σωστά. Όμως ε, η ερώτηση μου είναι εξής. Δεν τέλειωσε αυτή η προσπάθεια. Τι πιστεύετε ότι λείπει για να υπάρξει αυτό το θετικό τράνταγμα που είπατε, το θετικό σοκ για την οικονομία, ώστε οι πολιτικές και θεσμικές δομές της Ευρώπης να μην ε, καταρρεύσουν. Και ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για ένα πιο μακροπρόθεσμο όραμα για την ε, τετραπλής προεδρίας ε, καταγραφή και έκθεση. Τι νομίζετε ότι μπορεί να μας μπορεί να μας εξυπηρετήσει τώρα για να καθορίσουμε αυτό το όραμά μας για το μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Σας ευχαριστώ και όπως είπα προηγουμένως θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες μεταβλητές για να υπάρξει ανάπτυξη, καλές ευκαιρίες επενδυτικές και οικονομική πόρη. Νομίζω ότι το επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τεράστιο δυναμικό το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως και σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση των χρηματοοικονομικών πόρων για μόχλευση, αλλά και σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση ε, των επενδυτικών ευκαιριών. Και στο σημείο αυτό πιστεύω ότι υπάρχει θετική διάδραση μεταξύ των προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων στις χώρες και του νέου αυτού εργαλείου. Όπως μας υπενθυμίσατε, οι επενδύσεις μειώνονται. Και αυτό δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Επί σειρά ετών γίνεται αυτό. Και χρειαζόμαστε λοιπόν απελπισμένα επενδύσεις. Έτσι μεταφράζονται οι ευκαιρίες, οι επενδυτικές σε ανάπτυξη. Και αυτό μπορεί να γίνει λοιπόν έχοντας υπόψη και τα εθνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και αυτό είναι πολύ στο πνεύμα της νέας πρωτοβουλίας. Υπό το πνεύμα λοιπόν αυτό και από την οπτική γωνία αυτή πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει πιο έντονη διασύνδεση και αυτό ε, το προβλέπει το εργαλείο. Να συνδέσουμε λοιπόν τις επενδυτικές ευκαιρίες ε, και τις ε, ανάπτυξη γιατί η ενιαία αγορά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και αποτελεί τη μεγάλη μεταρρύθμιση στην οποία μπορούν να βελτιωθούν οι επενδύσεις. Θα πρέπει καλύτερα να κατανοήσουμε ποια είναι η σχέση μεταξύ ενιαίας αγοράς και των σχετικών πρωτοβουλειών και των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης. Αυτό συνδέεται δε ενδεχομένως με την μακροπρόθεσμη αυτή προπτική που αναφέρατε. Μακροπρόθεσμα πιστεύω ακράδαντα θα έλεγα ότι η Ευρώπη μπορεί να δώσει μεγάλη όθεση στην ανάπτυξη της καταργώντας τα εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ των χωρών, ε, επενδύοντας σε μεγάλες υποδομές, σε απτά κεφάλαια, στις τηλεπικοινωνίες, στην κοινοτομία. Πολλά μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να υπάρξει αυτή η νέα βάση καινοτομίας όπως ε, απονομάζεται. Αυτό και σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο προαπαιτεί συγκεκριμένη αξιοποίηση και κινητοποίηση των πόρων. Έχει έρθει λοιπόν ο χρόνος να το κάνουμε αυτό. Να υπάρξει αυτή η σύνδεση μεταξύ των νέων χρηματοοικονομικών μέσων, των επενδυτικών ευκαιριών, με τρόπο συνεργατικό. Τελευταία ευκαιρία επίσης να κατανοήσουμε πώς τα προγράμματα μεταρρύθμισης των χωρών μπορούν να έχουν επιρροή και στις άλλες χώρες, στις γειτονικές τους χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ, Λίγο ο Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής από το ECR, ο κύριος ε, Μαριάς. Ευχαριστώ, θα μιλήσω ελληνικά, Πρόεδρε. Κύριε Παντοάν, θεωρώ ότι η Ιταλική Προεδρία έδωσε μεγάλες υποσχέσεις, δημιούργησε προσδοκίες, αλλά δεν έφερε απτά αποτελέσματα, τα οποία να μπορούν να γίνουν αισθητά στην ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία. Ιδίως σε σχέση με το ζήτημα του δημοσίου χρέους, το οποίο δεν έχετε καν θίξει όπως επίσης δεν αντιμετωπίσατε την οικονομική καταστροφή, τη φτώχεια και την ανεργία που έχουν προκαλέσει στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου η λιτότητα, τα περίφημα προγράμματα προσαρμογής, τα μνημόνια. Και επειδή αναφερθήκατε στην Ελλάδα, ας δούμε τι έχει συμβεί εκεί. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή η πολιτική του μνημονίου και της Τρόικας έχει οδηγήσει σε ένα κοινωνικό αρμαγεδόνα. Παρότι η Ελλάδα έλαβε 215 δισεκατομμύρια ευρώ ως δάνεια από το 2010 μέχρι σήμερα ένα τεράστιο ποσό η ανεργία έχει φτάσει στο 26%. Η ανεργία των νέων στο 50%. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Έχουμε πάνω από 6 εκατομμύρια πληθυσμό, το 40%, που ζει σε κίνδυνο φτώχειας. Ταυτόχρονα, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ, αντί να μειωθεί με την πολιτική που αναφέρατε, αυξήθηκε από 120% του ΑΕΠ πριν το μνημόνιο και τη λιτότητα στο 180% του ΑΕΠ. Και όλα αυτά γιατί τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δουνουτού αντί να αξιοποιηθούν για να ενισχυθεί η πραγματική οικονομία, αντί να δοθούν στην πραγματική οικονομία, χρησιμοποιήθηκαν για να αναχρηματοδοτηθούν τα παλιά δάνεια. Επομένω απέτυχε κύριε Υπουργέ η πολιτική της Τρόικας στην Ελλάδα, η ευθύνη ανήκει στην Τρόικα που δημιούργησε αυτή την κατάσταση και εγώ έχω υποστηρίξει ότι εδώ χρειάζεται ένα σοκ, αλλά όχι αυτό που είπατε. Πρώτον, πρέπει να υπάρξει διαγραφή του επονίδης του χρέους. Πρέπει να αποζημιωθεί η Ελλάδα για την οικονομική ζημιά που έχει υποστεί από την πολιτική της Τρόικας πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φέτος να επιστρέψει 4 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι τα κέρδη που έβγαλε από τα ελληνικά ομόλογα τα οποία αγόρασε με έκπτωση 40% και τα πληρώνεται εις ολόκληρον. Αυτές είναι οι θέσεις δικές μου. Βεβαίως δεν πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε, αλλά θέλω να μας πείτε ποια είναι η θέση η δική σας για το κούρεμα του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα και στην Ιταλία που έχει φτάσει στο 135% και τελειώνω. Συμφωνείτε με τη σύγκληση ευρωπαϊκής διάσκεψης για το ευρωπαϊκό χρέος για να λύσει το θέμα του χρέους των Ευρωπαϊκών Νότο, να εφαρμόσει αυτά που εφαρμόστηκαν για τη Γερμανία το 1953 που κουρεύτηκε το χρέος της Γερμανίας 50% ήταν τα επιτόκια μηδενικά και το υπόλοιπο εξοφλήθηκε με ρήτρα ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Προσπαθώ να κατανοήσω ποια είναι η ερώτηση στη δήλωσή σας. Σε ό,τι αφορά την δήλωσή σας, ε, εξέφρασα ήδη τις απόψεις μου για την Ελλάδα, αλλά πιστεύω, αν σωστά κατανόησα και ζητώ συγγνώμη αν δεν κατάλαβα σωστά, αναφερθήκατε στο χρέος στην Ιταλία. Να σας πω το εξής λοιπόν, έχουμε μεγάλο χρέος. Το χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ του 2015, θα ξεκινήσει να μειώνεται από του χρόνου. Τούτου λεχθέντος, το ιταλικό χρέος είναι απόλυτα βιώσιμο. Μακροπρόθεσμα αναφέρεται από τους δείκτες βιωσιμότητας της, Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως από τα πλέον βιώσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως ε, χάρη στο σημαντικό, στη σημαντική μεταρρύθμιση του συνταξιβοτικού συστήματος που εισαγάγαμε σταδιακά τα τελευταία 10-15 χρόνια. Το Ιταλικό χρέος λοιπόν θα μειωθεί γρήγορα αν οι δυναμικές των τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στην Ευρωζώνη ήταν ε, κοντά στη φυσιολογική του τιμή, 2% δηλαδή, και οι διαστατικές μεταρρυθμίσεις επιπλέον που κάνουμε τώρα θα δώσουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Και αυτό πάλι θα συμβάλλει στη βιωσιμότητα. Αν η ερώτηση λοιπόν είναι ποια είναι η κατάσταση του Ιταλικού χρέους, αυτή είναι η απάντησή μου. Ευχαριστώ πολύ. For... Θα σε ευχαριστώ. Όχι. Ναι. Ναι, ναι. Α, σε δέκα δευτερόλεπτα μιλάει ο Πρόεδρος. Επόμενος. Ο μας απήντησε για το Ιταλικό χρέος. Σας ρώτησα και δεν απαντήσατε για το κούρεμα του ελληνικού χρέους. Η Ελλάδα πήρε όλα αυτά τα δάνεια και έχει γεμίσει ανέργους. Μόνο με κούρεμα του δημοσίου χρέους μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και προοπτική στη χώρα. Ευχαριστώ. Okay. Σας ευχαριστώ, αλλά πήρατε όλο το χρόνο. Αν είναι μεγάλη ερώτηση, δεν έχετε χρόνο για την απάντηση. Δεν απαντήθηκε το ερώτημα για το ελληνικό χρέος. Μάλιστα, επόμενος ομιλητής, η Κόρα Φανιουάζων από την ομάδα των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, Υπουργέ, που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω ευχαριστώντας και εσάς και την ομάδα σας για τη σκληρή δουλειά των τελευταίων έξι μηνών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θέμα του benchmarks, επειδή είμαι εισηγήτρια για το θέμα αυτό και διαπίστωσα τον τεράστιο όγκο δουλειά που κάνατε. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Να σας ρωτήσω λοιπόν για θέματα εφαρμογής των διευθυντικών μεταρρυθμίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειάζονται τόσο πολύ και για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, αλλά και για να βελτιωθεί η δημοσιονομική κατάσταση στα κρατημέλη. Δυστυχώς πολλά κρατημέλη δεν έχουν σημειώσει ιδιαίτερη πρόοδο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, των διθατικών αυτών μεταρρυθμίσεων. Μόνο 10% των συστάσεων αναχώρα κατά μέσο όρο εφαρμόζονται. Και πολύ φοβάμαι ότι για χώρες ε, όπως η Ιταλία και η Γαλλία αυτό το ποσοστό είναι πιο χαμηλό επειδή άκουσα την απάντησή στον συνάδελφο από το ΕΛΚ, αυτό δεν ε, ξέρω κατά πόσο είναι πολλά υποσχόμενα με την Ιταλία. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας, προτείνατε μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Μεγαλύτερη πίεση από τους ομοτήμους και μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη. Δεν συμφωνείτε ωστόσο ότι τα μέτρα αυτά είναι απίθανο να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και μπορεί να είναι και αντιπαραγωγικά. Δεν θα έπρεπε ανταυτού να επικεντρωθούμε στο πώς μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερα κίνητρα και μεγαλύτερες κυρώσεις για τα κράτη-μέλη. Προκειμένου το κατά πόσον τα κράτη-μέλη είναι ε, ενδεχομένως δικαιούχοι για ε, επιδοτήσεις να εξαρτάται από το κατά πόσον συνάδουν και συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας. Σας ευχαριστώ για απάντηση. Για τα καλά σας λόγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να αναφέρω τρία σημεία. Καταρχάς, μπορώ με σαφήνεια να σας πω ότι η ατζέντα της, ε, των διευθυντικών μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησής μου έχει επιταχύνει την, ε, τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων που κινούνταν ωστόσο προς την ίδια κατεύθυνση. Αναγνωρίζω, όπως είπα και προηγουμένως, ότι η χώρα αναγκάζεται να αντιμετωπίσει εμπόδια και προσκόμματα τα οποία δημιουργήθηκαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Άρα όχι μόνο περνάμε νόμους στο Κοινοβούλιο, αλλά φροντίζουμε να δίνουμε και τις εφαρμοστικές πράξεις για μεγάλες μεταρρυθμίσεις, ε, για την φορολογία, για το δικαστικό σώμα και το καθεξής. Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα για τις ε, διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις, αυτό συζητιέται ξανά και ξανά σε ό,τι αφορά τα θέματα πολιτικής. Η προσωπική μου άποψη για όσα μετράει είναι ότι δεν χρειάζονται τόσο μεγάλα κίνητρα σε ό,τι αφορά τα επιτόκια. Έχουμε χαμηλά επιτόκια στην χώρα μου, αλλά είμαστε σε ύφεση επί τρία χρόνια και θα πρέπει να αλλάξει αυτός ο ρούς και να δημιουργηθεί ανάπτυξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο προέρχεται από το ιστορικό της χώρας. Δεν χρειάζεται εξωτερική πίεση, εξωτερικά κίνητρα. Ένα άλλο σημείο, το τρίτο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ και το οποίο ενδεχομένως να είναι σχετικό για το μέλλον της κατάρτισης πολιτικής στην Ευρώπη είναι το γεγονός ότι ο αντίκτυπος οποιαδήποτε διαθετικής μεταρρύθμισης μεταξύ άλλων εξαρτάται από την κατάσταση των μακροοικονομικών συντελεστών. Υπάρχουν όλο και πιο πολλά στοιχεία μεταξύ άλλων και από το IMF και από τον ΑΣΑ ότι η μία αλλαγή μπορεί να έχει διαφορετικό αντίκτυπο ανάλογα με το κατά πόσον η οικονομία βρίσκεται σε κύκλο ανάπτυξη ή σε κύκλο ύφεση. Αν είναι ενδεχομένω να υπάρχουν καθυστερήσει. Και γιατί το λέω αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία ότι όλες τις χώρες θα πρέπει να κάνουν μεταρρυθμίσεις, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, ποιες είναι οι μακροοικονομικές ε, συνθήκες, σε ποια φάση του κύκλου βρίσκονται οι χώρες, γιατί, γιατί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να χρησιμοποιηθούν όλα τα μακροοικονομικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας η έννοια νομισματική πολιτική για την Ευρωζώνη και οποιαδήποτε άλλο περιθώριο έχουν οι χώρες στον προπολογισμό τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπάρμπαρα Σπινέλη από την Κουέτουρα. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Έχω δύο ερωτήσει. Μία για την Ευρώπη και μία για την Ιταλία. Ευρώπη. Σε λίγε εβδομάδε θα έχουμε εκλογέ στην Ελλάδα. Και εφόσον εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα, η Ευρώπη, συγγνώμη, θα πρέπει να λάβει επαναστατικέ αποφάσει περί λιτότητας. Τι θα γίνει λοιπόν με την ευρωπαϊκοποίηση του χρέους. Τι θα γίνει με τα χρέη της Γερμανίας από τον πόλεμο, από το 1953 η Ευρώπη πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που προτείνει ο Γιούγκερ. 20 δισεκατομμυριάκια που θα πρέπει να πάνε σε άλλους ε, προορισμούς με 300 δις δαπάνες μέσα σε τρία χρόνια και πώς θα γίνει αυτός ο πολλαπλασιασμός από το 1 στο 15. Όχι, θα πρέπει να υπάρξουν κρατικές επενδύσεις που να στηριχθούν από την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων με ευρωομόλογα. Και επίσης η ΕΚΤ με κρατικά ομόλογα διαφορετικής διάρκειας δεν θα πρέπει να παρέμβει. Θα ήθελα μια συγκεκριμένη απάντηση σε αυτές τις ελληνικές προτάσεις. Και για την Ιταλία. Δεν θα επιμείνω στους κανόνες περί ευελιξίας, αλλά τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους και δεν αρκεί να λέμε ευελιξία και η ευελιξία θα μας ε, έρθει αυτομάτως. Αυτό που μου φαίνεται πολύ σημαντικό στην Ιταλική πολιτική τώρα είναι η επίοικια που δείχνεται, που δείχνουμε ως προς τα δημοσιονομικά της χώρας με τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά να γίνονται εκτές και παρά τα τόσο ωραία ευρωπαϊκά μέτρα που έχουν εγκριθεί. Δεν θα παριθμίσω όλα τα άρθρα του τελευταίου νόμου της Ιταλίας που αποποινικοποιεί φορολογικά αδικήματα. Απλώς να θυμίσω ότι η η διαφθορά στην Ιταλία φέρνει μείωση 0,14% του ΑΕΠ. Και οι κανόνες περί διαφυγής είναι κανόνες που και εσείς είστε για την έγκρισή τους. Διότι και καταδικασμένοι για απάτη και φοροδιαφυγή όπως ο Μπερλουσκόνη έχουν διαφύγει. Και στις δύο περιπτώσεις, ακόμα και αν συμφωνείτε με αυτούς τους κανόνες ή τους αγνοούσατε, που είναι ίσως χειρότερο από τα δύο το δεύτερο, και στις δύο περιπτώσεις, τι απάντηση θα είχατε να μου δώσετε. Ευχαριστώ Υπουργέ. Thank you for your Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Κατά πρώτον, για τις προτάσεις και το τι θα προτείνει η μελλοντική ελληνική κυβέρνηση. Εγώ περιμένω πρώτα να τις δω. Μόλις έχουμε την ελληνική κυβέρνηση, η οποία πρέπει να εκλεγεί ε, με νόμιμες εκλογές, και αφού λάβει και ψήφο εμπιστοσύνη από τη Βουλή, τότε ω Υπουργό Οικονομικών μια χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα τοποθετηθώ και θα δω αυτέ τι προτάσει. Αλλά μου ζητάτε να σχολιάσω κάτι που είναι υποθετικό. Δεν το έχουμε ακόμα μπροστά μα, οπότε είναι αδύνατον να σχολιάσω. Ω προ τα σχόλιά σα για τα ιταλικά πράγματα, να πω τα εξή. Για να διευκρινίσω και σε αυτήν την ομάδα το τι συμβαίνει. Ο νόμος περί αυτό που αναφέρατε εσείς, ο νόμος φιναντσιάρια δεν περιέχει κανόνες, ούτε διατάξεις για την φοροδιαφυγή. Αυτό που εννοείται είναι η συζήτηση που ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη εντός του ονομαζόμενου ε, νόμου για τα φορολογικά που πέρασε από το Κοινοβούλιο το Μάρτιο του 2014 ο οποίος επιτρέπει στην κυβέρνηση να εγκρίνει δευτερογενή μέτρα για να βεβαιωθεί ότι το σύστημα των φορολογικών στη χώρα και οι εφορίες λειτουργούν τελείως αποτελεσματικά και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και για να μην υπάρχουν αβεβαιότητες για τους φορολογικούς νόμους. Μέρος αυτού του νομοσχεδίου συζητήθηκε από την κυβέρνηση στις 24 Δεκεμβρίου και μερικά από τα μέτρα που συζητήθηκαν από την κυβέρνηση ανεστάλησαν και αναπέμφθησαν στο κοινοβούλιο διότι θεωρήθηκε ότι υπήρχαν τεχνικά ψεγάδια σε αυτά τα κείμενα. Θεωρώ τον εαυτό μου μάλιστα υπεύθυνο για αυτά τα ψεγάδια και θα φροντίσω να διορθωθούν άμεσα. Θα τα δει λοιπόν πάλι η κυβέρνηση όλα αυτά και εφόσον τα εγκρίνει τότε θα σταλούν στο Κοινοβούλιο προς ε, ψήφιση. Δεν θα σχολιάσω λοιπόν τις ψευδεί κατηγορίες για την ε, εύνοια προς οποιοδήποτε συγκεκριμένο πρόσωπο. Απλώς τις αρνούμε κατηγορηματικά. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκίγκολ για τους πρασίνους. Welcome. Καλώς ήλθατε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνατε, κυρίως για την οδηγία για την νομοποίηση εσόδων παράνομες δραστηριότητες. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί και αυτό το έργο. Η Ιταλική Προεδρία έκανε πολλή δουλειά στον τομέα και έφερε τις διαπραγματεύσεις κοντά σε επιτυχές αποτέλεσμα. Κάτι όμως που δεν θα ολοκληρώσετε, δεν έχετε χρόνο, είναι ο τα τέλη των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Πώς θα συνδυαστεί αυτό με μέτρα για την φοροποφυγή και φοροδιαφυγή. Στις εφημερίδες ακούμε ότι στο θέμα των 11 υπάρχει κάποια κινητικότητα και θέλω να μου πείτε συγκεκριμένα. Συμφωνείτε ότι η φορολογική βάση πρέπει να διευρυνθεί και να μην περιλάβει μόνο μετοχές και παράγωγα επιμετοχών Μήπως θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα CDS παράγωγα δηλαδή επί του κρατικού χρέους. Δεύτερον, η αρχή της εντοπιότητας θα πρέπει να εφαρμοστεί και όχι μόνο ο τόπος της έκδοσης, αυτό λέει το Κοινοβουλίο και η Κομισιόν. Και τρίτον, δεσμεύεστε ότι ακόμη και αν ξεκινήσουμε με μια μεταβατική φάση, ότι θα δρομολογήσουμε και μια δεύτερη φάση, η οποία αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται με στόχο την ενοποίηση ακριβώς των φορολογικών βάσεων. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για τις ερωτήσεις σας. Όπως προείπα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της τελικής προεδρίας έγινε έργο με το G11 στο οποίο ανήκει βεβαίως και η Ιταλία Παρά το γεγονό ότι εγνώμαι δίσταντο, επί όλων των ζητημάτων που προναφέρεται, φορολογική βάση, αρχή φορολόγηση κλπ. Ε, και όχι τόσο προ την δεύτερη φάση, επ' αυτή ε, όλοι συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι είναι ανάγκη να προκύψει μια δεύτερη φάση. Ε, εν πάση περιπτώσει λοιπόν και παρόλα αυτά να σα πω ότι είχαμε εκτενεί συζητήσει και έχω την πεποίθηση ότι θα συνεχιστεί η σχετική συζήτηση με σκοπό να καταλήξουμε σε συμφωνία και προκειμένου να ευχαριστήσω όλους τους συναδελφούς, τους άλλους 10 δηλαδή του G11 που συνέβαλαν επικοδομητικά παρά τις διστάμενες απόψεις. Προσπαθήσαμε όλοι και προχωρήσαμε αργά αλλά σταθερά προς συμφωνία. Συγκεκριμένα τώρα, η Ιταλία καταρχήν είναι υπέρ της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης. Το ζήτημα είναι που θα σταματήσουμε. Αν θέσετε το ερώτημα σε κάθε μία από τις 11 χώρες, αν ρωτήσετε δηλαδή ποια είναι η απόψή σα σχετικά με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, θα πάρετε 11 διαφορετικές απαντήσεις. Δεν υπάρχουν καν τάσεις προς το παρόν μεταξύ των 11, αλλά πιστεύω ότι με περισσότερη προσπάθεια θα τα καταφέρουμε στο πρώτο ερώτημα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ναι, στην διεύρυνση, τη μέγιστη δυνατή διεύρυνση, αρκεί να καταλήξουμε στην κατηγορία αξιών που θα φορολογήσουμε. Δεύτερον, υπάρχει σχεδόν ένα φυσικό χάσμα μεταξύ μιας ομάδας, της ομάδας που ε, ασχολείται με το θέμα και που περιλαμβάνει και μεγάλες χώρες και μικρές χώρες. Οι δυνατότητες ε, διαφέρουν, καθώς και προτιμήσει μεταξύ μεγάλων και μικρών χωρών. Εξαρτάται το τι περιμένει να εισπράξει κάθε χώρα από κάθε διαφορετικό τρόπο φορολόγηση. Εγώ θα ήμουν υπέρ μιας προσέγγισης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη στον τόπο έκδοσης, σε κάποια άλλα μέτρα. Βεβαίω υπάρχουν τεχνικά μέτρα να συγκεράσουμε τις δύο προσεγγίσεις με την προπόθεση ότι όλα αυτά βεβαίω είναι εφαρμόσιμα, είναι εύκολα και που θα επιτρέψουν στις χώρες να έχουν κάποια επιπλέον έσοδα. Τέλος, και συγγνώμη για το αρχικό, τον αρχικό αλλά ναι, υπάρχει εν γέννη καταρχήν συμφωνία ότι πρέπει να υιοθετήσουμε μια βήμα προς διαδικασία ώστε να καλύψουμε όλων των ειδών τις αξίες και όχι μόνο όλες τις αξίες αλλά και άλλες χώρες πέραν δηλαδή των 11 Ευχαριστώ. Ο Μάρκο Τσάνι από το EFTD. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αφού άκουσα τα εισαγωγικά λόγια του Υπουργού Πάντων, μου φαίνεται σαν να έχω ζήσει τους τελευταίους έξι μήνες σε άλλο πλανήτη. Όλες αυτές τις επιτυχίες της Ιταλικής Προεδρίας εγώ δεν τις είδα. Κατά την άποψή μου ελάχιστα έγιναν στο επίπεδο της δουλειάς στο επίπεδο της φοροδιαφυγής ελάχιστα επίσης, εντάξει το τραπεζικό απόρριτο, αλλά το θέμα ότι η φοροδιαφυγή είναι εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι εξωτερικό με την περίπτωση του Λουξεμβούργου και άλλων κρατών όπως της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας, αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Την επιτυχία λοιπόν εγώ αυτή δεν την είδα. Και περνάω στις ερωτήσεις. Πρώτον, για τον απολογισμό του output gap, δηλαδή τις προσαρμογές στον προπολογισμό, στο διευθυντικό προπολογισμό, για τα χάσματα. Για το χάσμα παραγωγής λοιπόν, η Ιταλία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ε, πιστεύετε ότι πρέπει να υπολογίσουν αυτό το δίκτυο Ένα αποτέλεσμα για την αναθεώρηση της μεθοδολογίας υπολογισμού θα υπάρξει. Θεωρείται απειρχαιωμένη η, μεθοδολογία, η μέθοδος που προτείνεται. Υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον ΟΣΑ για τον ίδιο δίκτυο επίσης. Αυτό είναι μια απόδειξη. Δεν θα πρέπει να συστάθει αμέσως μια ομάδα εργασίας για να ξαναδεί αυτό αυτή τη μέθοδο που επηρεάζει τόσο πολύ ε, τα δημοσιονομικά των κρατών μελών και επίσης την άποψή σας για την ποσοτική χαλάρωση. Ε, κάτι που θα ξεκινήσει μάλλον από την ΕΚΤ. Θα υπάρξει κάποιος αντίκτυπος πραγματικά ή θα είναι ένα μέτρο που κατά την άποψή μου θα έχει μηδενικό αποτέλεσμα βλέποντας τα χαμηλά επιτόκια και τις ε, χαμηλότατους συντελεστές στα κρατικά ομόλογα. Βλέπουμε ότι όλα αυτά βρίσκονται στον αδύρ. Οι διαφορετικέ αλλαγές, διαφορές μεταξύ των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών των ΗΠΑ και της Ευρώπης είναι τεράστιες. Και Αύριο θα έχουμε ένα πρώτο κείμενο για το επενδυτικό πρόγραμμα Juncker. Εσεί μιλήσατε για επενδύσει, ανάκαμψη των επενδύσεων. Η ερώτησή μου είναι υπάρχουν καινούργια στοιχεία για το τι κατεύθυνση θα πάρουν οι επενδύσει, ακόμα και οι συγχρηματοδοτούμενες και πώς θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των ελλημάτων. Και βάσει των όσων ανακοινώθηκαν και από τα λόγια σας. Υποτίθεται ότι η Ιταλική Προεδρία έδωσε μάχη για τη μεγαλύτερη ευελιξία. Και έπειτα για την δουλειά που αναφέρατε, για, για την εργασία μάλλον στην Ιταλία, εγκρίθηκε νόμος για την ελαστικότητα, την ευελιξία. Όμως δεν χρειαζόμαστε την ευελιξία, δεν φέρνει η ευελιξία θέση εργασίας. Το ξέρετε πολύ καλά, διότι υπάρχει ένας δείκτης, ο δείκτης για την προστασία της εργασίας που έχει ετοιμάσει ο, ο ΣΑ. Με συγχωρείτε, αλλά σε 1,5 λεπτό θα σας δώσει τέσσερις απαντήσεις ο Υπουργός. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ. Try to be quick. Ε, θα είμαι σύντομος. Το χάσμα της παραγωγής. Εδώ Όντω, αυτό συζητήθηκε και στο Eurogroup και στο ECOFIN και είναι πολλέ οι χώρε που θεωρούν ότι η μέθοδο αυτή πρέπει να ανανεωθεί. Δεν έχω πολλά να πω για την ε, ποσοτική χαλάρωση και τι επιπτώσει τη δεν είμαι μέλος του Συμβουλίου της ΕΚΤ και το πώς θα καταρτιστεί αυτό δεν το ξέρω. Τώρα θα υπάρξει αντίκτυπο στην, γενικότερα στην αγορά και στον πληθωρισμό, το ελπίζω. Και εάν το πρόγραμμα Juncker θα συμπεριλάβει διαφορετικό υπολογισμό των επενδύσεων, δεν ξέρω. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ξέρω όσα και εσείς σήμερα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς όπως και για πολλά άλλα θέματα που τέθηκαν σε αυτή τη συζήτηση, αν είχα κάτι συγκεκριμένο να διαβάσω και να το σχολιάσω, θα έκανα, αλλά δεν το έχω τώρα. Ω προ την ευελιξία, εάν χρησιμοποιείτε για την δημιουργία θέσεων απασχόληση, αναφέρατε δίκτυ του όσα. Η δική μου αντίληψη για το θέμα είναι ότι η νομοθεσία για την προστασία της εργασίας είναι ένα από τα στοιχεία που επηρεάζουν και επηρεάζονται από την ευελιξία και τούμπαλιν ευελιξία χρειάζεται για να υπάρξει ανάπτυξη, για να υπάρξουν επενδύσει. Νομίζω ότι αυτά απαιτούνται για να υπάρξουν περισσότερε θέσει απασχόληση, συμπεριλαμβανομένε και τη χώρα μα. Ευχαριστούμε ο Μονό από του μη εγγεγραμμένου. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας το 2011 δηλώσατε ότι δεν πρέπει να αποκλείσουμε την πτώχευση κάποιων κατομέλων. Η χώρα σας, η Ιταλία, είδε τη βαθμολογία της από τη Standard Poor's να φτάνει το, το 2β. Εδώ ε, βλέπουμε ότι οι απαιτήσει των ομολόγων έχουν αλλάξει τελείως. Με τέτοιο χρέος σε 2.000, ε, σε 2.300 δις ε, σε σχέση με την Γαλλία ξεπερνάτε το χειρότερο μαθητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν τι δράσεις θα αναλάβετε. Δύο προτείνονται. Πρώτα απ' όλα οι μαζικές φιωτικοποίησεις. Ε, αναφέρατε ένα πρόγραμμα πωλήσεων στη χώρα σε 40% των εθνικών σιδηροδρόμων και του συστήματος εναέριου ελέγχου, εναέρειας κυκλοφορίας αλλά και στρατηγικά κομμάτια του κλάδου ενέργειας. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας, να στηρίξετε τις επενδύσεις, την ζήτηση, όχι. Θέλετε να σβήσετε το δημόσιο χρέος ε, μετά από τέσσερα χρόνια καθηγής διακυβέρνησης. Ως προς το χρέος λοιπόν βλέπω να ακολουθείτε την ίδια πορεία ε, με τη Γαλλία παρόλο που η Γαλλία δεν έχει και πολλά ακόμη να πουλήσει. Και επίση περισσότερο φεντεραλισμό στην Ευρώπη, αναθέτοντα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει τι απαραίτητε διευθυντικέ μεταρρυθμίσει. Με άλλα λόγια, μετά την απώλεια τη ε, δημοσιονομική και τραπεζική ε, αυτοκυριαρχία του, τα κράτη-μέλη θα χάσουν ε, και το δικαίωμα να ορίζουν την αγορά εργασία. Δηλαδή αυτά που είδαμε το Μάη του 68 στην Γαλλία αύριο θα γίνουν πραγματικότητα. Πώς θα γίνουν πράξη όλες αυτές οι οι μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι η ουσία του θέματος είναι να μείνει ο πυρήνας όλων το έθνος και να παραμένουμε στο εθνικό επίπεδο για του προπολογισμού παρά να υποκύπτουμε τα όσα ε, προκύπτουν ω κανόνε από την ΕΚΤ με το αμφισβητούμενο δικοπηλικό που προτείνεται ε, και την προσωπική χαλάρωση. Θα πρέπει να δούμε την χρηματοδότηση των εθνικών κεντρικών τραπεζών και να δοθεί ένα τέρμα στις ανοιχτές αγορές που έχει οδηγήσει σε πτώχευση κράτη όπως η Ελλάδα για παράδειγμα. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Thank you. Not... Σας ευχαριστώ. Δεν είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα τις ερωτήσεις, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω όπως και να έχει. Αναφερθήκατε στο πώς ε, αντιμετωπίζει η Ιταλία το πρόβλημα του χρέους. Είναι πρόβλημα αυτό, το αναγνώρισα. Αλλά νομίζω ότι αντιμετωπίζει το θέμα αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ξεφορτωθούμε το χρέος. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν είναι η ανάπτυξη. Και πάλι ανάπτυξη λοιπόν, η οποία ανάπτυξη όπως σας ανέφερα, επειδή δεκαετίας μειωνόταν. Να υπάρχουν λοιπόν ευκαιρίε ανάπτυξη και ευκαιρίε για θέσει εργασία και νομίζω ότι σημειώνουμε πρόοδο προ την κατεύθυνση αυτή. Άρα με πιο πολύ ανάπτυξη, το οποίο εξαρτάται πολύ, αλλά όχι πλήρω από τα δοτικά μέτρα τα οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση, θα υπάρξει πιο πολύ ανάπτυξη. Και αν καταφέρουμε να έχουμε πιο πολύ ονομαστική ανάπτυξη σε ό,τι αφορά την, ε, τον πληθωρισμό που είναι πέρα από τον έλεγχο των εθνικών κρατών θα έχουμε συνολική ανάπτυξη δεδομένων και των επιτοκίων των σημερινών και των ε, σημερινών προσπαθειών που διεξαγάγονται. Αυτό λοιπόν ήταν πάντα πρόβλημα επί σειρά δεκαετίων. Αυτό λοιπόν θα έβαζε στο σωστό δρόμο την Ιταλία. Επιπλέον υπάρχει ένα φιλόδοξο σχέδιο ιδιωτικοποίησης με δύο στόχους. Καταρχάς να συμβάλλει στη μείωση, στην ε, κατάργηση του χρέους και την μείωση του χρέους, αλλά και στην αύξηση πιέσεων ανταγωνιστικότητας ε, όπως ε, αναφέρατε στις εταιρείες που θα παραμείνουν στο δημόσια χέρια αλλά θα εκτεθούν σε πρακτικές διαχείρισης προκειμένου να υπάρχει καλύτερη αποτελεσματικότητα. Ύστερα, αναφερθήκατε στο ρόλο των εθνικών κρατών μελών, των κυρίαρχων κρατών μελών, σε σχέση με τις ευρωπαϊκές, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αναφερθήκατε στα θέματα των νομισματικών. Δεν θεωρώ την ερώτημα αυτό, θεωρώ την δήλωση. Δεν νομίζω ότι σας αναφέρω οποιοδήποτε μυστικό, δήλωνοντας ότι συμφωνώ με αυτά που υπονοεί η δήλωσή σας. Φυσικά λοιπόν χρειάζονται και τα εθνικά κυρίαρχα κρατημέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δύο ερωτήσεις και δύο απαντήσεις θα ακούμε από εδώ και πέρα. Τα Χούμπνερ και μετά Ρενάτο Σουαλβερ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, το Δεκέμβριο υπό την Προεδρία σας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε τη σημασία του πιο στενού συντονισμού της οικονομικής πολιτικής και συμφωνήθηκε ότι το Φεβρουάριο θα, αναλυτικό, θα υπήρχε ένα αναλυτικό σημείωμα και θα συζητιόταν αυτό στο άτυπο συμβούλιο και μετά θα προετοιμαζόταν ε, μια καινούρια έκθεση για το κατά πόσο θα συνεχιζόταν αυτό που έβαλε στο ράφι ο κύριος Φαρόμπαϊ. Δεν το ξέρουμε πλέον αυτό, ακόμα αυτό. Από αυτά που λέτε καταλαβαίνω ότι συμφωνείτε ότι χρειάζονται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για την βελτίωση της διαχείρισης της Ευρωζώνης. Και νομίζω ότι πολλοί συμφωνούν ότι είμαστε στη μέση μόνο των μεταρρυθμίσεων σε ό,τι αφορά θέματα διαχείρισης της Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει έλλειψη τεχνολογίας σε ό,τι αφορά τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις και καταλαβαίνω και εκτιμώ αυτό που κάνει η, Ευρωπα... η Ιταλία. Μιλάμε για ένα μόνιμο μηχανισμό, όχι για κάτι πρόσκαιρο και νομίζω ότι πολλοί συμφωνούν ότι έχουμε φτάσει στα όρια της τρέχουσας συνθήκης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη νομική βάση για κάποιες από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει προσφάτως. Δεν μας ικανοποιεί αυτή η βάση και φυσικά ξέρουμε ότι μπορούμε να τις βάζουμε από την πίσω πόρτα της μεγάλης μεταρρυθμίσης, αλλά αυτό συνήθως μας έρχεται μπούμεραν. Να ακούσουμε αυτό που είπε και ο κύριος Δράκη πρόσφατα. Είπε ότι η έλλειψη διευθυντικών μεταρρυθμίσεων οδηγεί σε αποκλήσεις μόνιμες στην Νομισματική Ένωση. Και αυτό φυσικά ε, δεν είναι καλό για κανέναν. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό η έλλειψη αυτού του μηχανισμού για αντραστικές μεταρρυθμίσεις. Ερωτώ λοιπόν στο πλαίσιο αυτό τι αναμένεται από την έκθεση της Προεδρίας σε ό,τι αφορά τις περαιτέρω μεταρρυθμίσεις της ε, διαχείρισης της Ευρωζώνης. Υπάρχει όρεξη για Μακροσκέλης μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε άλλη μια ερώτηση. Ο κύριος Ρενάτο Σόρου. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, και εγώ ήθελα να σας ευχαρώ για τη δουλειά σας, για τα τόσα αποτελέσματα που καταφέρατε και αναγνωρίστηκαν στην Ιταλική Προεδρία και σήμερα σε αυτή τη συζήτηση. Σήμερα το πρωί μαζί με άλλους συναδέλφους της Επιτροπής βρεθήκαμε στη Φραγκφούρτη, στην έδρα της ΕΚΤ και συναντήσαμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τα μέλη του Συμβουλίου της ΕΚΤ μας είπαν ότι οι νοσματικές πολιτικές από μόνες τους δεν φτάνουν, χρειάζονται και απαραίτητες δημοσιονομικές πολιτικές που θα πρέπει να υποστηρίζονται και από διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις όπως θυμήσατε οι οποίες έχουν επίδραση στι δημοσιονομικέ πολιτικέ και τι επενδύσει, δημιουργώντα το απαραίτητο επιχειρηματικό περιβάλλον ενδεχομένω για τι επενδύσει. Με ευνηδία όμω ένα από του ομιλωτέ λέγοντα ότι όλα θα ήταν πιο απλά εάν στην Ευρώπη είχαμε ένα σημαντικό ε, εργαλείο όπω τα ε, ευρωομόλογα. Και το σύγκρινε με άλλε γεωγραφικέ περιοχέ Είπε ότι Είναι πολύ δύσκολο να σκεφτούμε πως άλλες περιοχές το έχουν πετύχει και εμείς ως σύστημα όχι. Εγώ λοιπόν να κάνω μια αφελή ερώτηση. Τι χρειάζεται για να έχουμε ευρωμόλογα στην Ευρώπη. Καταλαβαίνω τα ιδιαίτερα εθνικά συμφέροντα, αλλά εντάξει υπάρχουν προσκεπτικιστές. Εμείς νομίζαμε ότι υπάρχει μια προοδευτική απογοήτευση με το ευρωπαϊκό εγχείρημα, αλλά με όσα συνέβησαν στη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες είδαμε μια αναπάντεχη απόκριση στην ε, σύγκληση όλων προς την Ευρώπη ε, και το είδαμε και πριν από λίγα λεπτά στην Ολομέλεια. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να σκεφτούμε ότι ενδεχομένως η Ευρώπη να χρειάζεται λίγο περισσότερο συνέστημα κάτι που να ξεπερνάει τις στιγμιαίες αντιδράσεις. Ίσως να τα δούμε αυτά με διαφορετικό βλέμμα και να βγούμε από αυτήν την ε, δύστιχη ύφεση και την ανεργία έχοντας μια διαφορετική προσέγγιση στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Πρόεδρος, πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και από τους δύο μιλητές. Ζητώ συγγνώμη αν δεν θα καταφέρω να απαντήσω ενδεχομένω πλήρω για το πρώτο σημείο που ακούσαμε, το θέμα της οικονομικής διακυβέρνηση. Είναι θέμα κλειδί και τώρα έχει έρθει ο καιρό να ξανασκεφτούμε την οικονομική διακυβέρνηση. Τώρα είναι ο όριμο το κλίμα γιατί δεν έχουμε βγει ακόμα από τη μεγάλη κρίση και ένα από τα παθήματα, τα, οποία, τα διδάγματα της κρίσης είναι ότι η Ευρώπη όχι μόνο θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη, ευέλικτη στην οικονομία της, αλλά να αναβαθμίσει τη διακυβέρνησή της για τις μελλοντικέ κρίσεις. Όλοι ξέρουμε ότι θα έχουμε και στο μέλλον κρίσεις. Μία σκέψη μόνο να προσθέσω στα αυτά που είπατε εσείς. Κάθε φορά που καταστρώνουμε εθνικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, να πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια εθνική διάσταση, αλλά υπάρχει και μια συστημική διάσταση. Με άλλα λόγια υπάρχουν στοιχεία τα οποία προαπαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση σε σχέση με την εθνική διάσταση και πάντα θα πρέπει να έχουμε υπόψη και τις δύο διαστάσεις. Και άρα ενδεχομένω, να συναγάγει κανείς ότι χρειαζόμαστε θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα πιο πολύ σε σχέση με τις συστημικές αυτές ε, προκλήσεις. Το δεύτερο σημείο, η αφελής ερώτηση είναι πάρα πολύ επίκαιρη τα ευρωομόλογα και φυσικά με τα ευρωομόλογα εννοούνται πολλά και διαφορετικά εργαλεία για πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς, ωστόσο με ένα κοινό στοιχείο πάντα. Πρόκειται για ένα θέμα χρέους, σε ό,τι αφορά εκδότη χρέους, ο οποίος είναι η Ευρώπη. Για να συμφωνήσουμε λοιπόν σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο χρέους έναντι των επενδυτών, θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή τοποθέτηση. Και αυτό σχετίζεται με το συστημικό θέμα που μόλις έθεσα. Πρόκειται για ένα θέμα κοινή ε, αξιοπιστής, αν θέλετε. Κοινή θεώρηση των προβλημάτων σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του χρέους, ε, διευκόλυνση της ε, προσαρμογής. Αυτό είναι ο ευρωπαϊκός, η ευρωπαϊκή διάσταση. Για να υπάρξει όμως αυτό θα πρέπει να υπάρχει κοινό στόχος, κοινή αντίληψη. Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο το οποίο εξ ορισμού θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκό. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Τελευταία δύο ερωτήματα. Ο κύριος Μαρτουσέλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αναγγείλατε ότι το 2015 το δημόσιο χρέος της Ιταλίας θα αυξηθεί για ένα μεγάλο μέρος της χρονιάς και θα υπάρξει περικοπή των δαπανών με αύξηση των επιτοκίων. Με την εξοικονόμηση που προγραμματίζεται 30 δισεκατομμυρίων πιστεύετε ότι ούτως ή άλλως θα αυξηθεί το χρέος ή χρειάζονται προς τα μέτρα. Και πώς θα δοθεί η όθηση στις επενδύσεις με τα προγράμματα που υποτίθεται θα χρηματοδοτηθούν από την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπάρχει κάποια εκδήλωση, κάποια, κάποια ένδειξη ενδιαφέροντος από την, ε, και κάποιες ειδήσει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η κυρία Μπερές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αναφέρατε τις ε, οικονομικές συνθήκες που αντιμετώπισε η χώρα σας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Έχω την εντύπωση ότι δεν μιλήσαμε τόσο πολύ για μια διάσταση που ήταν απροσδόκητη με την ε, ύφεση στον θεσμό και την ε, απασχόληση ήταν η πτώση των τιμών του πετρελαίου. Αυτό είναι καλό. Δεν το λέμε τόσο πολύ και όμως έχει σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και για να τα πω τα πράγματα λίγο ομά, το όφελος από την ε, πτώση στις τιμές του πετρελαίου να τα αφήσουμε στην ε, αγορά να το διαχειριστεί ελεύθερα δεν υπάρχει τρόπος να αξιοποιήσουμε την πτώση των τιμών για να Ε, δημιουργήσουμε ένα νέο πόρο, μια νέα πηγή που θα μπορούσε να στηρίξει τις επενδύσεις, βλέποντας προσπάθειες που έχουν γίνει και σε άλλους καιρούς. Με μηχανισμούς προσαρμογής, με την απόσπαση νέων πόρων. Και μετά μιλήσατε για τις προκλήσεις ε, τι επικοινωνιακέ που μα αναμένουν από αύριο στα πλαίσια τη συζήτηση για την απελεξία, πώ βλέπετε την προετοιμασία και τη συνέχιση τη Προεδρία σα. Διότι επί τη ουσία μπορούμε να φανταστούμε ότι οι συζητήσει για την οικονομική διακυβέρνηση ε, ξεκίνησαν στην δική σα Προεδρία απλώ, αλλά το χρονοδιάγραμμα θα επεκταθεί. Πώ βλέπετε το κείμενο περί που θα εκδοθεί αύριο τέλος πάντων αύριο ή μεθαύριο θα λάβουμε γνώση και την έκθεση των τεσσάρων προεδριών βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμη ένα κενό εδώ ε, ένα περιθώριο για πράγματα που θα μπορούσαν επιπλέον να γίνουν Πώς θα διεξαχθεί η συζήτηση λοιπόν για την οικονομική διακυβέρνηση εγώ θα περιμένουμε τη μεγάλη βραδιά των ε, τεσσάρων προέδρων και τι περιμένετε να υπάρχει στην ανακοίνωση που θα μας γνωστοποιηθεί αύριο μεθαύριο Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για το ευρύτερο φάσμα των ερωτήσεων για το θέμα του χρέους. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυβέρνησης μας, το 2015 θα αυξηθεί η αναλογία χρέους ως προς το ΑΕΠ. θα πέσει από το επόμενο έτος και αυτό είναι άσχετο με τις διαδικασίες για την ειδικοτικοποίηση. Αυτό έχει να κάνει με τη δυναμική του ΑΕΠ και του πληθωρισμού των τιμών. Για το δεδομένο οικοδόμημα των επιτοκίων. Αυτό λοιπόν, οι ιδιωτικοποίησεις θα αυξήσουν την ιδιωτικοποίηση του χρέους. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε να επιταχύνει την χρηματοδότηση επενδύσεων, δεδομένου ότι υπάρχουν πόροι και ότι υπάρχουν και νέα project. Αναφέρθηκα στην Task Force για τα επενδυτικά προγράμματα που δημιουργήθηκε Έχουμε λοιπόν νέα project τα οποία θα μπορούσε να εξετάσει η ΕΤΕΠ και αυτό γίνεται από ό,τι γνωρίζω. Έχουμε λοιπόν εργαλεία στην Ευρώπη για να δώσουμε όθηση στην ανάπτυξη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για ερωτήσεις για τις συνολικές τιμές. Σε ό,τι αφορά τις τιμές του πετρελαίου. Αυτό ασφαλώς θα επηρεάσει τις ε, αγορές και αυτό θα αξιοποιηθεί ιδιωτικά εκτός αν υπάρχει spillover και ωφελήσει αυτό και τον προϋπολογισμό αυτό επαφείται στα νοικοκυριά στις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά το τι θα κάνουν αυτές το γνωρίζουν καλύτερα σε ό,τι αφορά τα ωφέλη για τον προϋπολογισμό υπάρχει πιο πολύ δημοσιονομικός ε, χώρος και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπο φιλικό προς την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόληση. Τι θα πρέπει να κάνουμε για την ευελιξία. Θα δούμε τι θα πει αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά ανεξαρτήτως αυτού θεωρώ ότι η ευελιξία δεν αποτελεί αυτό σκόπο. Είναι κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ενισχύσουμε την δημιουργία ανάπτυξη και θέσεων απασχόληση. Θα πρέπει να ενταχθεί λοιπόν στη στρατηγική συζήτηση που ελπίζω ότι θα λάβει χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Πάντων, τον Ιταλική Προεδρία και όλους τους συνεργάτες και αξιωματούχους της Ιταλικής Προεδρίας που εργάστηκαν τόσο σκληρά για να στηρίξουν την νομοθετική εργασία και δουλειά που τόσο πολύ σχολιάσαμε. Νομίζω ότι το εξάμενο ήταν ιδιαίτερα καρποφόρο και ακόμη και αυτή η ανταλλαγή απόψε με τον Υπουργό Πάντοαν ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστούμε και πάλι τον Υπουργό Πάντοαν και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία με την ε, Ιταλική κυβέρνηση για τις προκλήσεις των ερχόμενων μηνών. Let's... Συνάδελφοι, Επόμενο σημείο στη μερική διάταξη ακρόαση με τον Στέφαν Κόφερερ αναπληρωτή γενικό γραμματέα του ΟΣΑ Καλώς ήλθατε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ Θα συζητήσουμε την επισκόπηση του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης διαπιστώσει και προκλήσεις. Εξαιρετικά επίκαιρο το ζήτημα. Έχουμε ήδη στα χέρια μας το κείμενο από την εισηγήτρια και αύριο περιμένουμε την ανακοίνωση περί ευελιξίας. Το θέμα που ήδη συζήτησαμε με τον Υπουργό, τον κύριο Παντοάν. Συζητήσαμε τις προκλήσεις, την έκθεση των τεσσάρων πρόεδρων, τη βελτίωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, την ανακοίνωση του Μηχανισμού Συντονισμού των Ευρωπαϊκών Οικονομικών Πολιτικών παρούς συνθήκες αναγκαίες αλλαγές ένα σωρό δηλαδή ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε ξεκινώντας όμως από τι πρέπει να κάνουμε στην παρούσα συγκυρία το σύμφωνο σταθερότητας δηλαδή περιμένουμε κάτι από την Κομισιόν αύριο Περιμένουμε κάποιες εξελίξεις, σημαντικές εξελίξεις που με τη σειρά μας θα συζητήσουμε. Οπότε, είμαι βέβαιος ότι η συζήτηση είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Δίνω μέσω τον λόγο στον κύριο Κάφερερ για 10 λεπτά θα κάνει μια εισαγωγική παρατήρηση και εν συνεχεία θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις για την εισηγήτρια και την ομάδα διαπραγμάτευσης. Και εάν μας μείνει χρόνος θα ακολουθεί ένα τύπου eye διάστημα ερωτήσεων και απαντήσεων. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, βουλευτές, είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι εδώ σήμερα. Ξέρω ότι ήταν δύσκολη η μέρα σας. Άκουσα για συναντήσεις ε, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γνωρίζω για την συζήτηση με έναν προκατοχό μου. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, ο κύριος ε, δούλευε για τον ΩΣΑ προηγουμένως, πριν να γίνει δηλαδή υπουργό Οικονομικών Οικονομίας και Οικονομικών Υποθέσεων της Ιταλίας. Είναι μεγάλη λοιπόν τιμή για μένα, παραλαμβάνω, που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων άκουσα κάποιον ρωτάει ποιο είναι το σωστό μείγμα πειθαρχία και ευελιξία στο ευρώ. Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε ισορροπία μεταξύ διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, δημοσιονομικής πολιτικής και νομισματικής πολιτικής. Όμως η συζήτηση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Επιτροπή σας είμαι βέβαιος καθώς προβαίνουμε σε μια επισκόπηση της κατάστασης βάσει και της έκθεσης ε, το ερώτημα είναι πώς συγκεράζονται όλα αυτά τα τρία. Το δεύτερο είναι ότι οι συνθήκες αλλάζουν, οπότε και η σωστή ισορροπία διαφέρει. Σήμερα από αυτήν που θα με προκρίνει πριν από δύο-τρία χρόνια. Και σίγουρα σε 2-3 χρόνια από τώρα πάλι οι συνθήκε θα έχουν μεταξύ αλλάξει και θα είναι διαφορετικέ από τι σημερινέ. Οπότε πάλι θα πρέπει να προκρίνουμε το σωστό μείγμα, τη σωστή ισορροπία τη στιγμή εκείνη. Ένας άλλος λόγος για ότι νομισματική δημοσιονομική πολιτική και διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσεις είναι ένα μείγμα το οποίο αλλάζει, είναι ότι σε κάθε τομέα η πρόταση είναι διαφορετική. Ας πούμε, στην δημοσιονομική εξυγένση έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε πολλές χώρες. Κάποιοι θα πούνε βεβαίω όχι αρκετοί, όμως όλοι γνωρίζουμε ότι οι λόγοι χρέους ΑΕΠ μειώθηκαν από το ως το 2014 έχουν μειωθεί κατά 2,5% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη και έχουμε και ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο μειώθηκε πρώτος δηλαδή και στη δημοσιονομική πολιτική και αυτό το οποίο έχουμε σήμερα είναι το ερώτημα τι θα γίνει με την νομισματική πολιτική εγώ θα πω δύο λόγια επί δύο βασικά ζητημάτων το πρώτο είναι Υπάρχει αρκετή ευελιξία στο πλαίσιο της σημερινής κατάστασης, όπου αντιμετωπίζουμε δηλαδή υψηλή ανεργία σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ, μα πολύ χαμηλό πληθωρισμό. Πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε πολλές από τις χώρες μας και παρόλα αυτά τελματωμένη παραγωγή. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, μήπως σε αυτήν την συγκυρία που υπάρχει κίνδυνο τερμάτωση τη οικονομία, ε, υπάρχει περίπτωση να χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία. Επ' αυτού λοιπόν θα μιλήσω και θα πω και δύο λόγια για το τι πρέπει να κάνουμε με το τέλος αυτής της κατάστασης. Όταν επανέλθουμε δηλαδή σε κανονικές οικονομικές συνθήκες στην Ευρωζώνη όπως ίσχυε άλλωστε για δεκαετίες και ελπίζω σύντομα να συμβεί και πάλι αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση, βρισκόμαστε στο αναπτυξιακό ή ηφαισιακό μέρος του κύκλου, του οικονομικού κύκλου. Αν ρίξετε μια ματιά στο κείμενο της Κομισιόν, με σίγουρο ότι το διαβάσετε, είναι σαφές ότι υπάρχει περιθώριο ευελιξίας για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε προβλήματα στο θερικό μέρος του κύκλου. Αλλά αυτό είναι πολύ μικρό περιθώριο ευελιξίας. Αν ερμηνεύσουμε τους υφισταμένους κανόνες με τρόπο μηχανικό, επαναλαμβάνω είναι βέβαιο ότι η ευελιξία είναι ελάχιστη και ότι οι δυνατότητες ποσοτικής απελευθέρωσης είναι πολύ μικρές. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ρεαλιστική προσέγγιση. Αυτό αναζητήσαμε και τα τελευταία δύο χρόνια και τι κάναμε. Διευρύναμε, παρατείναμε τις προθεσμίες για τη συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια. Ξέρετε ότι αυτή η ευελιξία χρησιμοποιήθηκε 11 φορές τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό ήταν που μπορούσαμε να κάνουμε στο πλαίσιο μιας ρεαλιστικής προσέγγισης. Λίγη όμως ευελιξία, περιορισμένη ευελιξία. Εμείς ως όσα πιστεύουμε ότι σαφώς η συγκυρία είναι εξαιρετική ασυνήθιστη να δούμε τα επιτόκια της ΕΚΤ είναι μια συγκυρία στην οποία χρειαζόμαστε τόνωση της οικονομίας για μας λοιπόν έλεγα ότι είναι σαφές ότι σήμερα και αύριο θα χρειαστούμε δημοσιονομική στήριξη της ζήτησης Πρέπει μας όλες οι κυβερνήσεις να εμπλακούν, να επιδοθούν σε σοβαρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Έγιναν σαφώς πολλές, αλλά χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερες για να μπορέσουμε να τονώσουμε μακροπρόθεσμα την ζήτηση στην Ευρωζώνη. Με βάση αυτήν την πεποίθηση γνωρίζουμε ότι θα χρειαστούν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στη σημερινή έκτακτη συγκύρια εξαιρετική συγκυρία. Πιστεύουμε ότι η Ευρωζώνη πρέπει να είναι πιο επεκτατική όσον αφορά τη δημοσιονομική της πολιτική. Και αυτό μπορεί να γίνει με αποφάσεις του Συμβουλίου. Να ξέρουμε δηλαδή να υπάρχει βεβαιότητα ότι δεν θα τιμωρηθούν ε, κάποιες χώρες εάν λάβουν τη μία την άλλη πρωτοβουλία. Κύριε Πρόεδρε, μόλις είπατε ότι θα συζητήσουμε το σχέδιο Αύριο συγκεκριμένα πιστεύουμε ότι ο μηχανισμός του σχεδίου Juncker πρέπει να επιτρέπει ενισχύσεις των επενδύσεων του ε, σχεδίου. Αυτό πρέπει να είναι απολύτω σαφέ για να τονώσουμε τη ζήτηση. Μετά, τι θα κάνουμε όταν τελειώσει η κρίση. Θα χρειαστούμε και άλλες μεταρρυθμίσεις, άλλες αλλαγές των δημοσιονομικών κανόνων που ισχύουν σήμερα. Με προκειμένου έχω πω τρία πράγματα για τα, μετά την κρίση. Πρώτον, πιστεύουμε στον ΩΣΑ ότι ένας εξορπημένος προπολισμός είναι πολύ σημαντικός βεβαίως στο πλαίσιο του συμφώνου όμως όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα όταν έχετε η να προβούμε σε διαπιστώσεις και να κάνουμε προβλέψεις Πρέπει να δούμε λοιπόν την διαρθρωτική κατάσταση ξεχωριστά από χώρα σε χώρα για να βρούμε τη σωστή απάντηση. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί παρατηρητές, να βρούμε σε αξιολογήσεις πολύ προσεκτικά γιατί εξής της έλλειψης αυτών αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Ο Πάντουα έλεγε στις εφημερίδες πριν από λίγες μέρες ότι η Κομισιόν και ο ΣΑ καταλήγουν σε διαφορετικά νούμερα, σε διαφορετικές αξιολογίες, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προβούμε κοινή αποτύπωση της κατάστασης. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις πρέπει η μεθοδολογία να επανεξεταστεί Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πιο σοβαρά τις κατατόπους συνθήκες όταν μετρούμε το χάσμα της παραγωγής, το output gap, καθώς και την τάση της ανάπτυξης. Αυτά θα είναι όλο και πιο σημαντικά στο μέλλον. Δεύτερη πτυχή, δεύτερο ζήτημα που θέλω να τονίσω είναι τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια χαριστοποιείται το με την οικονομία. Και εδώ η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η προσπάθεια της εξυγίανσης είναι διαφορετική φύση από χώρα σε χώρα και εκεί πρέπει να βοηθήσουμε τα επόμενα χρόνια. Κάποιες ε, χώρες δημιούργησαν, ίδρυσαν εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια για να μπορέσουν να πετύχουν εξορροπήση των δημοσιονομικών τους και αυτό είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Και τρίτον, η πολυπλοκότητα του δημοσιονομικού πλαισίου στην Ευρωζώνη. Αν ρωτήσετε τον απλοπολίτη τι ξέρετε για το δημοσιονομικό πλαίσιο και τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωζώνη, οι περισσότεροι ίσως ενδεχομένως θυμηθούν το περίφημο 3% του ελλείμματος του προπολογισμού. Και αυτό δεν είναι παράδοξο, διότι είναι κάτι το οποίο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς. Όμως όλοι γνωρίζουμε σε αυτήν την αίθουσα ότι υπάρχουν και άλλοι στόχοι και άλλοι κανόνες ανάλογα του πλαίσιο. Υπάρχει το η διαθετική εξορρόπηση του προπολογισμού, υπάρχουν τα χρέη, υπάρχουν άλλα κείμενα και κανόνες, πράγματα τα οποία πολύ δύσκολα καταλαβαίνει ο απλό άνθρωπος. Και να μην πω ότι και οι κυβερνήσει ελάχιστα καταλαβαίνουν, διότι οι κυβερνήσει προσπαθούν μάλλον να δουν πώς θα αξιοποιήσουν του κανόνε για να του υπερκεράσουν για να ξεφύγουν ακριβώς από αυτούς τους κανόνες. Εμείς στον ΩΣΑ είμαστε πεπισμένοι ότι χρειάζεται να απλουστευτεί το πλαίσιο αυτό και από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβάλλουμε στην προσπάθεια αυτή. Απλούστευση, δηλαδή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητός. Έχουμε τον κανόνα του χρέους. Έχουμε τους μεσοπρόθεσμους στόχους. Έχουμε το περίφημο 60% και έχουμε και τον μεσοπρόθεσμο στόχο όμως για τις περισσότερες χώρες. Εδώ ισχύουν δύο κανόνες, δύο διαφορετικοί κανόνες για το ίδιο θέμα, Άλλο με τη χώρα. Λοιπόν, επειδή περνάει η ώρα, να που εγκατακλείδει το ΩΣΑ συνεργάζεται στενά με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κομισιόν υπέρ των μεταρρυθμίσεων. Κάναμε σημαντικό έργο στην αποτίμηση των επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων. Παρακολουθούμε τις νομισματικές μεταρρυθμίσεις διότι εμείς έχουμε κάθε λόγο ως οργανισμός μαζί με πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και στο μέλλον για να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εννοείται στο μέλλον κάθε φορά που θα χρειαστεί να αναθεωρήσουν για άλλη μια φορά το δημοσιονομικό πλαίσιο. Πιστεύω ότι όλοι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι σίγουρα θα χρειαστεί μια άλλη μια διαφορετική αναθεώρηση στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω σε μια επικοδομητική συζήτηση. Σα ευχαριστούμε πολύ Στέφαν. Κάπφερε, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση και δίνω το λόγο στην Περπάς που είναι η συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση. Πρέπει να πω ότι δεν περίμενα απαραίτητο να συγκλίνεται τόσο πολύ με τι δικέ μα τι απόψει. Αλλά χαίρομαι διότι αυτά που είπατε εδώ απόψε επιτρέπουν να τροφοδοτήσουμε την μελέτη της όλης δουλειάς που έχουμε καθορίσει. Υπάρχει όμως ένα σημείο αφετηρίας. Κάτι καθοριστικό. Είπατε ότι υπάρχει θέμα σωστής ισορροπίας, οπότε πρέπει να δούμε σε τι πλαίσιο κινούμαστε. Και για αυτή τη σωστή ισορροπία μιλήσατε για την νομισματική, τη δημοσιονομική πολιτική και τις διαδοτικές μεταρρυθμίσεις. Εάν δούμε όμω την ετήσια εξετασία ανάπτυξη όπω την παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφήνει κατά μέρο την νομισματική πολιτική. Και προσθέτουν ένα τρίτο πυλώνα, ε, μια τρίτη κορυφή του τριγώνου, τι επενδύσει. Εσεί το θέμα των επενδύσεων το εξετάζετε σαν συνέπεια ε, μετά από τη διαπίστωσή σα για το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή Όντω στη διάρθρωση αυτή των διαφορετικών σημείων προ μελέτη δεν είναι ε, το όλο ζητούμενο οι επενδύσεις. Δεν έχουμε έρθει σε μια τέτοια διαρθρωτική κατάσταση όπου υπάρχει έλλειψη επενδύσεων, υποεπενδύσεις. Ε, οι συγκυρίες είναι τέτοιες, έχουν υποβαθμιστεί τα δημοσιονομικά και τα κράτη-μέλη δεν κάνουν αυτά που έπρεπε. Αλλά ίσως δεν είχαμε και τους κατάλληλους κανόνες για να βεβαιωθούμε ότι έχουμε μια ε, βέλτιστη κατάσταση για τις επενδύσεις εντός Ευρωζώνης. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη αφορά το περιθώριο εγκλημών μας ε, με τους υπάρχοντες κανόνες. Είπατε ότι είναι λίγοι και ότι είστε ανοιχτός προκειμένου να συζητηθεί η αναθεώρησή τους, το, η δέσμη αυτή δημοσιονομικών κανόνων. Επί της ουσίας δηλαδή, μεγάλο περιθώριο σημαίνει ότι δεν υπάρχει αρκετό, μπορούσε να υπάρξει και λίγο παραπάνω. Άρα έχουμε περιθώριο λοιπόν. Και τρίτη ερώτηση, για να αφήσω και άλλους συνάδελφους να λάβουν το λόγο, για τα κράτη-μέλη και τις διαρθρωτικές τους μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι σε μια διαπίστωση συμφωνούμε όλοι. Οι μεταρρυθμίσεις ε, είναι ένα πράγμα αλλά δεν ε, πρέπει να συγχαίρεται με το βαθμό προστασία που προσφέρει η συμμετοχή στην Ευρωζώνη. Και άλλο πράγμα είναι η συνειδητοποίηση και ανήλυψη ευθύνη από τα κράτη-μέλη για τι διεθνωτικέ μεταρρυθμίσει. Δεν πιστεύετε ότι σήμερα η Τρόικα, η, η, η ποιότερη Τρόικα, που θα μπορούσε να είναι βάση συμφωνία, δεν είναι αντιπαραγωγική ω προ την ανάληψη ευθύνη για αυτέ τι ε, διορθωτικέ μεταρρυθμίσει. Και μια τελευταία παρατήρηση. Αναφέρατε το Ανώτατο Συμβούλιο των Δημοσιονομικών, ε, λέγοντας ότι έχουν παίξει καλό ρόλο σε πολλά Δεν θα έπρεπε προς συμφέρον όλων και για να έχουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή συζήτηση για τα κίνητρα, τις ανισότητες μεταξύ κρατών, τη σωστή διάγνωση για την Ευρώπη. Δεν θα έπρεπε να γίνει μια δικτυωμένη συζήτηση αυτού του Συμβουλίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να φωτιστεί σωστά η ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος με την εμπειρογνωμοσύνη τους που έχει περιοριστεί μόνο σε μερικα κάτι κράτη-μέλη για την ώρα. Ευχαριστώ, παρακαλώ. Κύριε Καπφέρε. Ευχαριστώ, κύριε Συγγετρία. Θα προσπαθήσω να απαντήσω εν συντομία και συγκεκριμένα στα ερωτήματα που θέσατε. Καταρχάς, ναι, ο ΣΑ είναι πεπισμένος ότι χρειαζόμαστε πιο πολλές επενδύσεις. Το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2015 θα επικεντρωθεί ακριβώς στις επενδύσεις. Αλλά είναι πολύ σαφέ ότι οι επενδύσει δεν είναι μόνο δημόσια φύση και είναι σαφέ επίση ότι δεν πρόκειται μόνο για θέμα διαχείριση τη ζήτηση, αλλά και θέμα διαχείριση τη προσφορά. Πιστεύουμε επίσης ότι εξετάζοντα τον κανονισμό του δημοσιονομικού πλαισίου υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με μια πολιτική φιλική προς τις επενδύσεις. Δυνατότητα για παράδειγμα μακροπρόθεσμης προοπτικής αν οι μεταρρυθμίσεις έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την, το κλίμα το επενδυτικό. Αυτό σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να οργανώνεται με, τρόπο φιλικό προς τις επενδύσεις, αλλά ότι υπάρχουν κάποιες ιδέες στον κανονισμό που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να είναι φιλικές προς τις επενδύσεις. Περιθώριο ελιγμό. Ελιγμού είπατε, ναι. Όπως είπα πριν, ναι, στην τρέχουσα κατάσταση θα πρέπει να σκεφτούμε μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών. Αλλά από την άλλη η αξιοπιστία είναι εξίσου σημαντική όπως και το περιθώριο ελιγμού. Αυτό που είδαμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια είναι το εξή. Κάποιες χώρες μέλη στην Ευρωζώνη, στην, Ευρωπαϊκή, στην Ευρωζώνη χάσαν αξιοπιστία γιατί είχαν πιο πολύ χρόνο να οργανώσουν τις μεταρρυθμίσεις, τις διαστατικές μεταρρυθμίσεις και να αντιμετωπίσουν το έλλειμμα. Και μετά από κάποια χρόνια τελικά όχι μόνο εφαρμόστηκαν όλες αυτές οι διαστατικές μεταρρυθμίσεις, αν δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, χρειάζονται και σαφής δέσμευση, σαφής αξιοπιστία για τις μεταρρυθμίσεις αυτές τις διαρθωτικές. Συμφωνώ ότι το να συζητήσουμε την ιδιοκτησία των... σε ποιον ανήκουν τελικά αυτές οι διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις είναι πολύ σημαντικό. Η Ευρώπη τελικά είναι αυτή. Να σας υπενθυμίσω ότι ο ΣΑ πέρσι τον Νοέμβριο κατήρτασε ένα έγγραφο για την γαλλική κυβέρνηση προσπαθώντας να υπολογίσει τον αντίκτυπο των ε, διαθετικών μεταρρυθμίσεων στη Γαλλία προκειμένου να υποστηρίξει αυτές τις διαθετικές μεταρρυθμίσεις για τη γαλλική κυβέρνηση. Αλλά στην τελική ανάλυση είναι σαφές ότι είναι πολύ καλύτερο να είναι εθνικής ε, προέλευσης αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πτυχή για να διοργανωθεί συνεργασία μεταξύ των εθνικών συμβουλίων δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Τα εθνικά συμβούλια υπάρχουν και σε πολλές ευρωπαϊκές, ευρωπαϊκά ζητήματα, όπως για παράδειγμα για τη μείωση του γραφειοκρατικού άχθους, της ε, γραφειοκρατίας. Ξέρω ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ, για παράδειγμα, εμπειρογνωμόνων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας. Ξέρω λοιπόν ότι είναι κάτι το ευπρόσδεκτο η συνεργασία των Εθνικών Συμβουλίων. Κανείς δεν πρόκειται να αντιταχθεί. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Να ζητήσω από τους συναδέλφους και από τον ε, καλεσμένο μας να τηρήσουν ε, τον κανόνα των χρονικών ήρων των 5 λεπτών. Η Έστα Ντελάν είναι η επόμενη από το ΕΛΚ. Δεν είναι εδώ. Μα τη βλέπω πουθενά. Ο Μπέντ Λούκε λοιπόν από το ECR, από τους Ευρωπαίους ε, Μεταρρυθμιστές και Συντηρητικούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ερωτήσω για την ε, υπόθεση, την, θέση ότι χρειαζόμαστε πιο πολύ ευελιξία. Τα ασφάλματα της ιστορίας ε, δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται. Αλλά το έχουμε ζήσει ξανά στην Ευρωζώνη αυτό το θέμα και για την ε, μεγαλύτερη ευελιξία το 2005 και αυτό τροφοδότησε σε μια μεγάλη κρίση από την οποία δεν έχουμε εξελθεί ακόμα. Το κρατικό, το δημόσιο χρέο είναι μεγαλύτερο από ποτέ και τώρα πάλι ζητάτε μεγαλύτερη ευελιξία παρά το γεγονός ότι αυτά που είχαμε συμφωνήσει ως τώρα ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν. Τα ελλείμματα και τα όρια του ελλείμματος πάντα παραβιάζονταν θέμα του ισοσκελισμού της, ε, του προπολογισμού δεν τηρείται σχεδόν από κανένα, παρόλο που ορίζεται από τη συνθήκη. Μιλώντας λοιπόν για την ευελιξία, πάντα μιλάμε για μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες. Αυτό θέλουμε να δικαιολογήσουμε. Γιατί στους πολιτικούς σε εποχές κρίσεων, τίποτα δεν το πιο πολύ από το να υπάρχουν μεγαλύτερε δαπάνε, για να υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική κίνηση. Από πού ξέρετε όμως, πώς ξέρετε ότι η κρίση οφείλεται σε μειωμένη ζήτηση. Μήπως έχουμε πρόβλημα ανταγωνισμού στην Ευρωζώνη. Μήπως δεν υπάρχει επένδυση γιατί δεν είναι ανταγωνιστικές οι επενδύσεις στην Ευρωζώνη. Γιατί τα προϊόντα που ξερετε ομω πω ξερετε οτι η κριση οφειλεται σε μειωμενη ζητηση μηπως εχουμε προβλημα ανταγωνισμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πολλούνται παγκοσμίω γιατι τα προιοντα που παραγονται υπάρχουν καλύτερε και πιο ευνοϊκέ τιμέ. υπάρχουν πιο ανταγωνιστικές ε, μέθοδοι παραγωγή. Πού ξέρετε σίγουρα ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση αν υπάρχει άλλο πρόβλημα ουσιαστικά, το θέμα του ανταγωνισμού. Αν θέλετε λοιπόν να τονώσετε τις επενδύσεις, πείτε μου πού θέλετε να τις τονώσετε. Ο οικονομολόγος θα έλεγε εκεί που είναι μεγαλύτερη η παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα της επένδυσης. Ρωτώ λοιπόν, η παραγωγικότητα των επενδύσεων είναι πιο υψηλή στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία ή στη Γερμανία, στις κατοχώρες, στη Γαλλία. Πού θέλετε να γίνουν επενδύσεις. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό. thank you, Mr. for Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, κύριε Λουκέ. Έχετε δίκιο. Η κρίση του 2005 των κανόνων μας. Ήταν μια δυσάρεστη εμπειρία. Όλοι πλέον συμφωνούμε ότι ναι μεν χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία αλλά δεν είναι μόνο ευκαιρία η ευελιξία είναι και απειλή. Είναι επίσης σαφές ότι η συζήτηση περί περισσότερης ευελιξίας δεν ε, εξώνεται μόνο με υψηλότερες δημόσιες δαπάνες. Και το θέμα δεν είναι και πάλι η έλλειψη εναγωνιστικότητας κάποιων βιομηχανιών διεθνώς. Ίσα ίσα που κάποιες βιομηχανίες στην Ευρώπη είναι πολύ ανταγωνιστικές. Τις ξέρουμε. Ίσα ίσα μάλιστα που ακριβώς λόγω της αύξησης των μισθών και περιοριστήρων σε κάποιες ασιατικές χώρες η βιομηχανική παραγωγή σε ορισμένους τομείς επιστρέφει στην Ευρώπη. Αυτό το βλέπουμε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Ε, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα σε διάφορες χώρες της Ευρωζώνης. Φυσικά δεν φτάσαμε στο τέλος, δεν πετύχαμε αυτά που θέλαμε, αλλά δεν τα πάμε και τόσο άσχημα στον τομέα της ανταγωνιστικότητας. Πού θα επενδύσουμε, είπατε. Βεβαίω. Καταρχήν, δεν μιλάμε μόνο για δημόσιου πόρους. Το σχέδιο Juncker βασίζεται εν μέρη σε δημόσιε επενδύσει, αλλά αποτελεί ενθάρρυνση και σε ιδιωτικές επενδύσεις για να έχουμε ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Συμφωνώ λοιπόν ότι πρέπει να επενδύσουμε εκεί όπου θα έχουμε την υψηλότερη απόδοση, να επενδύσουμε με επιχειρηματικά κριτήρια αλλά όχι μόνο στην Ολλανδία και την Φιλανδία. Πρέπει να έχουμε παρουσία και σε χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Δείτε ας πούμε την κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Η διασύνδεση Γαλλίας-Ισπανίας είπαμε σίγουρα θα τονώσει, θα βοηθήσει την ενιαία αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Αυτό θα βοηθήσει την Ευρώπη, θα είναι καλό για τις επιχειρήσεις στην Ισπανία, για τις επιχειρήσεις στη Γαλλία σίγουρα θα πάρουμε τα λεφτά μας πίσω. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ο μηχανισμός Connecting Europe ενάντια στην Ευρώπη, διασύνδεση στην Ευρώπη, χάρη στις υψηλής ταχύτητας συνδέσεις στο διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αυτό κάνει αυτή τη στιγμή, αναζητά λοιπόν ευκαιρίες επένδυσης στις οποίες θα επενδύσουμε τόσο δημόσια κεφάλαια, κρατικά κεφάλαια, όσο και ιδιωτικά. Κύριε Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αναπληρωτά, Γενική Γραμματέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτησή σας, την παρέμβασή σας. Θα ήθελα σε γενικό επίπεδο, από το γενικό επίπεδο μάλλον, να περάσω στο επίπεδο της λεπτομέρειας και να θέσω κάποια ερωτήματα. Για παράδειγμα, έχουμε την εξής κατάσταση στην Ελλάδα, όπου συζητιέται κατά πόσον θα υπάρξει κούρεμα, κατά πόσον χρειάζεται απαλλαγή από το χρέος, όπου το θέμα της ευελιξίας και της οικονομικής, ε, των οικονομικών κινήτρων και το ποιος θα πρέπει να διαθέσει τα, α, τις πιστώσεις, ε, δημιουργούν βάσιμους φόρους ότι μεγαλύτερη ευελιξία θα σημαίνει σε ε, υποχώρηση των διευθυντικών αλλαγών στην Ελλάδα. Πώς ε, αξιολογείται τις ε, συστάσεις του ΩΣΑ σε σχέση και με χώρες όπως η Γαλλία ή όπως η Ιταλία που δεν είναι υπό το κόθεστος διάσωσης και όπου ο τα τελευταία χρόνια έχει εκδώσει συγκεκριμένες συστάσεις Ρώτησα για την κυρία Πάντοβα το κατά πόσο εφαρμόζονται αυτές οι συστάσεις που εκδίδει ο Θα ήθελα λοιπόν να θέσω πιο συγκεκριμένο το ερώτημα αυτό. Πιστεύετε ότι η ευέλιξη, ευέλικτη αυτή διαμόρφωση των κανόνων που αναφέρατε είναι αντιπαραγωγική για τις κυβερνήσεις, γιατί οι κυβερνήσεις πάντα δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να εξηγήσουν στους πολίτες την αναγκαιότητα της διευθυντικών αλλαγών. Πιστεύετε λοιπόν ότι από πλευρά του ΩΣΑ υπάρχει κάποια σύσταση για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί και να εφαρμοστεί καλύτερα οι διευθυντικές αυτές αλλαγές. Για να είμαστε, για να είμαι κύριε αυτά που συζητήσαμε έως τώρα δεν αποτελεί εναλλακτική για τις ε, χώρες του μνημονίου σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις από τα άλλα κρατημέλη του Συμφώνου σταθερότητα. Και αυτό σημαίνει ότι είναι σαφές ότι όταν μιλάμε για δημοσιονομική ευελιξία δεν μιλάμε για τις καταστάσεις, για τις περιπτώσεις αυτές. Μιλάμε για το νομικό πλαίσιο για όλα τα κρατημέλη της Ευρωζώνης. Μιλώντας για τις συστάσεις για τα, τις χώρες του Μνημονίου, ο ΣΑ μπορεί να εκδώσει μόνο συστάσεις για τα κράτη-μέλη ή για τους εταίρους μας. Το τι κάνουν από εκεί και πέρα είναι απόφαση των εθνικών κυβερνήσεων, είναι σαφές. Αλλά αν με ρωτάτε, είμαι βέβαιος ότι για παράδειγμα όταν κοιτάμε τη διαδικασία ιδιωτικοποίηση, ακόμα πολλά πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα. Υπάρχει ακόμα σύσταση του ΟΣΑ για την ιδιωτικοποίηση στην Ελλάδα, την είναι απαραίτητη και αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια δεν αποτελούν επαρκή πρόοδο από πλευρά δική μα, αλλά αυτό είναι σαφέ ότι επαφείται στα χέρια τη εθνική κυβέρνηση και όλοι ξέρουμε ότι οι εκλογέ θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ρόνια Ικάρη από την ΚΟΕ τώρα. Ευχαριστώ και να σας ευχαριστήσω για την εισαγωγική σας παρουσίαση. Ε, να σας θυμίσω δικές σας μελέτες που έχουν δείξει ότι υπάρχει εντυνόμενη ανισότητα, αυξανόμενη ανισότητα στις χώρες του ΩΣΑ. Η κρίση έχει πλήξει τα φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού. Και μάλιστα πολύ σοβαρά. Αλλά δεν είναι εκείνοι που θα αποφεληθούν αν υπάρξει ανάκαμψη. Οπότε και πλήττονται περισσότερο από την κρίση και δεν ωφελούνται από την ανάκαμψη. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη όξυνση των ανισοτήτων. Εμποδίζει την ανάπτυξη και εμποδίζει την πρόοδο της κοινωνίας όπου υπάρχει ένταση των ανισοτήτων. Ενώ εμείς θέλουμε να μειώσουμε τις ανισότητες στην κοινωνία. Εφόσον λοιπόν μεταρρυθμίζουμε την οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να δούμε και τους δείκτες που πρέπει να συμπεριλάβουμε για να καλύψουμε τις ανισότητες. Έχω τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις βάσει του στόχου να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες. Τι δείκτες πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν ε, θέλουμε να αξιολογήσουμε τα κάτι μέλη στην ετήσια αξιολόγηση των οικονομιών τους και πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε τις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις. Πώς μπορούμε να προβλέψουμε το αν θα περιορίσουν τις ανισότητες στην κοινωνία ή όχι. Και τρίτον, συμφωνείτε μαζί μου ότι αν συνεχίσουμε στην πορεία που τώρα έχουμε λάβει, διαρκώς θα εντείνονται οι ανισότητες. Κάτι που βλάπτει γενικώ στην κοινωνία μας. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας σε αυτή τη συζήτηση και την όλη μελέτη του θέματος. Ευχαριστώ. Έχετε δίκιο. Το θέμα των ανισοτήτων στις κοινωνίες μας είναι ένα ζήτημα προτεραιότητας για τον ΩΣΑ. Η... Το τελευταίο έγγραφο εργασία μας το αναφέρει. Δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο, όπως είπατε. Μήνυμα των έγγραφου αυτού ήταν ε, όχι απλώς ότι οι ανισότητες αυξάνονται από δεκαετίες σε πολλές χώρες του ΩΣΑ, αλλά ότι υπάρχουν ε, στοιχεία για το ότι οι υπερβολικές ανισότητες ε, αποτελούν φραγμό για την ανάπτυξη στις χώρες μας. Δεν είναι λοιπόν θέμα ηθικό ή δεοντολογικό ή πόση ανισότητα θέλουμε ή δεν θέλουμε. Ε, ανισότητες θα υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες, είναι δεδομένο, αλλά αυτό που μας απασχόλησε ήταν τι μπορούμε να κάνουμε για να προωθήσουμε την ανάπτυξη τη κοινωνία μας. Και μία από τις πτυχές που πρέπει να καλύψουμε είναι η... ο αναχαιτισμός των ανισοτήτων. Οι συστάσεις, οι πολιτικές συστάσεις που θα βρείτε σε αυτό το έγγραφο είναι ο βασικός λόγος που η αύξηση των ανισοτήτων ε, ταυτίζεται με την παρεμπόδιση της ανάπτυξης τη χώρα αυτές. Γιατί, Γιατί τα χαμηλότερα εισοδήματα επενδύουν λιγότερα στην εκπαίδευση, για τα, λιγότερο στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Οπότε δεν μιλάμε για αναδιανομή όταν θέλει κανείς λόγω χάρη να επενδύσει περισσότερο στο εκπαιδευτικό σύστημα τη στήριξη των φτωχότερων τμήματων του πληθυσμού. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι αυτή η ανάπτυξη που δεν λαμβάνει η χώρα οδηγεί σε υποβάθμιση της εκπαίδευσης στην όλη διαδικασία ε, και ιδίω για τα φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού και αυτό είναι το πρώτο μας πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν απαντώντας την ερώτηση θα πω εάν, ε, ότι είναι δύσκολο να σας απαντήσω για το αν η εν εξέλιξη μεταρρυθμίσει μπορούν να περιορίσουν τι ανισότητε. Βραχυπρόθεσμα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Κάποιε δεν ξέρουμε αν θα έχουν τέτοιο αποτέλεσμα. Η μεταρρύθμιση όμω του εκπαιδευτικού συστήματο ε, ελπίζουμε να βελτιώσουν την κατάσταση στα κρατη και την διάσταση της ισότητας. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε έτσι συνολικά ότι κάθε διαφορετική μεταρρύθμιση οδηγεί σε περισσότερες ανισότητες της χώρας μας. Δεν ευσταθεί αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε η ο κύριος Ούρτασον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Θα ήθελα δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις να σας κάνω. Πολύ με ενδιαφέρει η έκθεση για τις προοπτικές απασχόλησης του 2014 που παρουσιάσατε στο ΩΣΑ και ιδιαίτερα για ένα από τα στοιχεία και τις συστάσεις για την οικονομική πολιτική αναφέρατε στις μεταρρυθμίσεις ότι μία από τις διορθωτικές μεταρρυθμίσεις και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μείωση των μισθών είχε πάει υπερβολικά μακριά σε κάποιες περιπτώσεις και ότι αυτό επηρεάζει σε κάποιες περιπτώσεις κεντρωμένες περιοχές την ε, ανάκαμψη. Θα μπορούσατε να υπησέλθετε σε λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά αυτή την ιδέα που παρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, έτους αυτού και πιστεύετε ότι η μισθή και η μείωση των μισθών σε κάποιες περιφερειακές ε, περιοχές είναι σε τόσο χαμηλό επίπεδο, σε τόσο υψηλό επίπεδο μάλλον η μείωση που είναι αντιπαραγωγική. Κάτι άλλο τώρα που θα μας βοηθούσε ιδιαίτερα στην δουλειά μας. Συμφωνώ ότι τα κρατή-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται περιθώριο ελιγμού για τα δημοσιονομικά του στο παρόν στην τρέξουσα συγκυρία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αν εφαρμοστού η ευελιξία, πιστεύετε ότι επαρκούν οι τρέχοντες κανόνες ή χρειάζεται μεταρρύθμιση προκειμένου σε μια κατάσταση όπως η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να έχουν τους μηχανισμούς που χρειάζονται προκειμένου να αντιδρούν όπως θεωρούν ότι χρειάζεται. Η απάντηση. Ξέρετε ότι ο Σά είναι πεπισμένος ότι οι καλοπληρωμένες δουλειές χρειάζονται. Χρειάζονται στα κράτη-μέλη μας και γι' αυτό για παράδειγμα, προτείνει τη Γερμανία, στη Γερμανία όσοι, όσα στην τελευταία έκθεση να υπάρξει κατώτατος μισθός στη Γερμανία. Ναι, όντως υπερβολικά χαμηλοί μισθή μπορεί να έχουν αντίκτυπο και στη ζήτηση. Είναι σαφές αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις σε χώρες του μνημονίου για τη μείωση των δημοσίων δαπανών για το εργατικό δυναμικό στον δημόσιο κλάδο, για παράδειγμα, ήταν εσφαλμένες. Όταν συγκρίνουμε τους δημοσίους υπαλλήλου, το σώμα των δημοσίων υπαλλήλων σε διάφορες χώρες του ΩΣΑ, θα διαπιστώσετε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πολύ, μεγάλη, πολύ μεγάλες ε, διαφορές και υπάρχουν υπερτροφική δημόσιοι κλάδη και εκεί λοιπόν θα πρέπει να μειώσουμε τους δημόσιους, ε, τις δημόσιες δαπάνες ε, είτε μειώνοντας τους μισθούς είτε μειώνοντας το εργατικό, μειώνοντας το εργατικό δυναμικό. Αυτό είναι πρόβλημα ζήτησης. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε αυτόματα ότι είναι θέμα ζήτησης. Γιατί αν είναι υπερβολικά υψηλές οι δημόσιες δαπάνες για το δημόσιο κλάδο υπάρχουν υπερβολικά λίγα χρήματα μετά για άλλους κλάδους όπως η εκπαίδευση. Άρα θα πρέπει να υπάρχει σωστή ισορροπία. Ευχαριστώ πολύ ο Μάρκο Βάλλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε για το θέμα των ανισοτήτων και επειδή βλέπουμε ότι συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια ο πλούτος, σε λίγες μέρες θα υπάρξει μια συνάντηση, μια νέα συνάντηση του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ και θα συζητηθεί και το θέμα αυτό. Τελευταία, βλέπουμε λοιπόν συγκέντρωση του πλούτου στις χρηματοπιστωτικές αγορές, εις βάρος της πραγματικής οικονομίας, ιδίως στην Ευρωζώνη. Οπότε, πού μας οδηγεί αυτό σε προβλήματα του αποπληθωρισμού, ότι το χρήμα δεν κυκλοφορεί στην πραγματική οικονομία, στις τσέπες των πολιτών. Και πέρσι το ανέφεραν πολλοί οικονομολόγοι, είπαν ότι πολλές χώρες της Ευρωζώνης ε, βρισκόνται στα πρόθυρα του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, που έχουν ένα μέτρο ελάχι, ελάχιστου εισοδήματο και στήριξής του. Υπάρχει λοιπόν ένα περιθώριο στις συνομιλίες σας για να αποφύγουμε λίγο την αποπληθωρισμό. Αυτό το παράδεκτο φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού να μην γίνει καθεστώς στην Ευρώπη. Πρέπει να δώσουμε χώρο στις ε, υποκρίσεις χώρες ώστε το πλούτο που μπορεί να αποσπάσουν να τον προσφέρουν σε αυτή την στήριξη του του εισοδήματος και με την ανάκαμψη της οικονομίας είδαμε ότι το να δίνει κανείς χρήμα στις χρηματοδοτικές αγορές δεν ε, δίνει κανένα αποτέλεσμα και είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι θα συνεχίσει να μην υπάρχει αλλαγή έτσι. Νομίζω είναι σαφές αυτή την αποφάση των εθνικών ε, κυβερνήσεων. Εκείνοι πρέπει να σκεφτούν ε, τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας σε κάθε χώρα και όταν μιλάτε για τις ανισότητες, εάν δείτε την έκθεσή μας, Επικεντρώνονται στις ανισότητες στις επιμέρους χώρες. Όχι στην ανισότητα μεταξύ χωρών η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, και αυτό είναι και το ενδιαφέρον, έχει αμβλύνει τις ανισότητες μεταξύ χωρών. Και αυτό είναι χρήσιμο να το γνωρίζουμε στη συζήτηση. Και άλλη μια πτυχή, ίσως να έχετε δίκιο, 5-6 χρόνια πριν, Πολλέ ήταν οι επενδύσει στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ, αλλά ξέρουμε ότι αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Τι βλέπουμε να γίνεται τώρα, ε, περισσότερε επενδύσει στα πραγματικά ενεργητικά, στην πραγματική οικονομία. σω μεσοπρόθεσμα να υπάρξει και εδώ πρόβλημα αν δημιουργηθεί σαπουνόφουσκα. Έχει συμβεί σε κάποιε χώρε τη Ευρωζώνη. Όμω προ στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ το χρήμα στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ. Στα πραγματικά ενεργητικά το βλέπουμε. Uh, Ευχαριστούμε. Και τώρα λίγος χρόνος για Catch the Eye. Δύο ομιλητές έχω. Τον κύριο Ροζάτη και μετά την κυρία Φερέιρα. Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα επενδύσεων στην Ευρώπη, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών. Οι δημόσιες επενδύσεις συρρυκνώνονται λόγω δημοσιονομικών περιορισμών. Οι ιδιωτικές δεν πρόκειται να προκύψουν σύντομα λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης και λόγω της αβεβαιότητα των προοπτικών της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και λόγω του υψηλού χρέους. Στις προτάσεις Υπάρχει κάτι για την απομείωση του χρέους επιχειρήσεων και νοικοκυριών, κάτι το οποίο θα, τις, θα τους επιτρέψει να αυξήσουν τις ταπάνες τους για να τονωθεί η ζήτηση. Ή τελειώς πώς θα επιβιώσουμε με τόσο υψηλά επίπεδα χρέους. Δεν πρόκειται ποτέ να αυξηθεί η ζήτηση στην Ευρώπη. Και δεν, δεν θα έρθει βεβαίως έτσι και η ανάπτυξη. Να ομοδοποιήσουμε την πρώτη με τη δεύτερη ερώτηση. Ελίζα, παρακαλώ. Δεύτερη ερώτηση, ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν εξαιρετικά χρήσιμη παρουσία σας, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά το χάσμα της παραγωγής και το πρόβλημα του υπολογισμού του και πώς υπολογίζουμε και τα διαρθρωτικά ελλείμματα κλπ. Ξέρουμε από μελέτες του ΩΣΑ ότι έχετε μια εικόνα της κατάστασης αλλά θέλω να μου πείτε εσείς τι έχετε να πείτε για το θέμα της ευελιξίας και των κυρώσεων και ότι όλα αυτά στηρίχθηκαν σε ελλειπείς μετρήσεις, σε ελαττωματικές μετρήσεις. Δηλαδή βλέπουμε ξαφνικά και η Κομισιόν, ακόμα και Κομισιόν από το προς στην Άνοιξη αλλάζει τους υπολογισμούς της. Εδώ θα υπάρχει θέμα αξιοπιστίας της διαδικασίας μετρήσεων των στατιστικών. Ύστερα όλοι μας λέμε ότι πρέπει να ακολουθούνται οι προτάσεις, πρέπει να γίνονται οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά πρέπει να αναλύουμε και τις προτάσεις τις συστάσεις. Γιατί κάποιες χώρες <laughs> ακολούθησαν τις συστάσεις και βρέθηκαν εν μέσω μιας τρομερής ύφεσης και δεν μπορούν να βγουν με τίποτα. Και τέλος, μια ερώτηση για το μέλλον. Είμαστε μια, σε μια νομισματική ένωση. Η σύγκληση δεν θα έρθει χάρη σε κάποιο το χέρι. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη αναζήτηση λύσεων, ίσως και στο πλαίσιο της έκθεσης των τεσσάρων πρόεδρων. Λοιπόν, θα γίνει κάποια συζήτηση. Πώς θα συγκεράσουμε όλα τα συμπεράσματα βάσει των διαγνώσεων που κάνετε κι εσείς. Για να μάθουμε κάτι περισσότερο έστω σχετικά με το μέλλον μας. Ευχαριστώ. Πρώτο ερώτημα. Επενδύσεις και πάλι. Είπατε να επιταχύνουμε τη μείωση του χρέους για να προκύψουν κονδύλια και επενδύσεις. Ίσως κάποιοι συναδελφοί σας μάλιστα να υποστηρίξουν ότι α ας επενδύσουμε πρώτα και μειώνουμε μετά το χρέος. Γι' αυτό ακριβώ. Απόψε συζητούμε το σωστό μήμα, το σωστό συνδυασμό μεταξύ ευελιξίας, αξιοπιστίας, πλαίσιο κλπ. Πιστεύω ότι το πρώτο είναι η εξουπιστία στις χρηματοοικονομικές αγορές. Γιατί πολλές φορές αυτή η εξοπιστία δεν προκύπτει από τις δημόσιες επενδύσεις. Εξαρτάται και από τις, ή μάλλον επηρεάζει και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Γιατί οι επενδυτές είναι στην Κίνα, στις ΗΠΑ, στην Ινδία, παντού. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι χρειαζόμαστε πρώτα εμπιστοσύνη, να υπάρχει εμπιστοσύνη στις μεταρρυθμίσεις μας, να είμαστε αξιόπιστοι ω προς τις μεταρρυθμίσεις μας. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος και έτσι θα τονώσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις. Φυσικά, αν μειώσουμε το έλλειμμα μας σε μηδέν όπω έγινε στην Γερμανία πέρσι, θα λέω στη Γερμανία συγκεκριμένα ότι δεν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω επενδύσεων, αλλού πρέπει να γίνουν επενδύσει. Τώρα, τι επενδύσει αυτέ τι περιμένουμε από το σχέδιο Juncker. Ξέρουμε βεβαίω ότι μέσω πρόθεσμα τουλάχιστον το σχέδιο Juncker δεν είναι αρκετό παρά την μείωση, την πτώση της τιμής του πετρελαίου παγκοσμίως. Είναι και αυτό αρκετό όμως όχι. Γι' αυτό λέω άλλη συζήτηση για τα μεσοπρόθεσμα και, άλλο, και άλλη για τα, για τα βραχυπρόθεσμα και άλλη για τα μεσοπρόθεσμα. Κύριε Φεραίρα, αναφέρετε πάρα πολλά στις ερωτήσεις σας. Θίξατε πολλά ζητήματα, δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να τα απαντήσω όλα. Θα χρειαζόμαστε μια ολόκληρη συνεδρίαση. Αλλά είπατε για την ύφεση σε κάποιες χώρες λόγω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Όχι, είναι ποικίλη κατάσταση που χώρα σε χώρα. Δείτε την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία. Εκεί θα δείτε ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. Βέβαια, από πλευρά αναπτυξιακή τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα στην Ελλάδα, αλλά εν τέλει το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει άμεσο συσχετισμό ευθεία σχέση μεταξύ μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι οι διαθροτικές μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητε για να, ως προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη στο μέλλον. Είπατε επίσης για κυρώσεις και για την βεβαιότητα και τις μεγάλες διακυμάνσει στην οικονομία των χωρών μας. Εμείς υποστηρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή στην παρούσα συγκύρια χρειάζεται περισσότερη ευελιξία ακριβώ λόγω της αβεβαιότητας στις χώρες μας. Είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί κατά επανάληψη στη στη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς ήμασταν υπέρ της ευελιξίας, δεν, έχει, δεν πέτυχαμε να πείσουμε. Και η συζήτηση υπέστρεψε στις κυρώσεις. Τώρα, για το δημοσιονομικό πλαίσιο και πάλι, η σύστασή μας είναι απλούστευση. Αυτό το είπατε και εσείς, ε, κυρία εισηγητρία στην έκθεσή σας. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Εγώ ήμουν Υφυπουργό Οικονομικών στη Γερμανία πριν χρόνια, ίσως να το θυμάστε αυτό, και θυμάμαι πολύ καλά όλε τι συζητήσει που είχαμε στα εθνικά κοινοβούλια, με τι εθνικέ κυβερνήσει σχετικά με το αναθεωρημένο δημοσιονομικό πλαίσιο, σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμεινο και όλου του νέου κανόνε που τότε θεσπίσαμε. Για του πολιτικούς και τα κοινοβούλια το ξέρω, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο να πλουστεύσουν τις διαδικασίε. Όμω, αν θέλουμε να ενστερνιστούμε τις αλλαγέ αυτές και να γίνουμε πιο αξιόπιστοι, αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε αποτελέσματα, τώρα δεν υπάρχει άλλο δρόμος. Πρέπει να πλουστεύσουμε τι διαδικασίε. Φιλόδοξο ο στόχο, αλλά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτά, ευχαριστώ όλοι πρόεδρο. Για ένα γρήγορο σχόλιο, λοιπόν, τελική παρατήρηση, το λόγο δεν είναι στην εισηγήτρια. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχουμε ήδη αρχίσει. Ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, πραγματικά. Υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία μπορούμε να επανέλθουμε, αλλά θα τα κάνουμε και σε τεμερέ επίπεδο. Κάποια σχόλια για την τελευταία παρατήρηση. Το πρώτο σχόλιο. Για την επένδυση που θα πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά την ανάλυση για το χάσμα παραγωγής. Εδώ ενδεχομένω να υπάρχει ε, περιθώριο ελιγμού για κάποια ευελιξία. Αλλά επί της ουσίας η ανάλυση σας μας οδηγεί στο να διαπιστώσουμε ότι το χάσμα παραγωγής δεν είναι κάτι το σταθερό. Πώς μπορεί λοιπόν να υπάρχει κάποιο συμπέρασμα βάσει στοιχείων που είναι τόσο δύσκολο να τα επεξεργαστούμε. Το πρόβλημα, όπως λέτε, είναι ότι δεν εφαρμόζονται οι κυρώσεις. Ναι. Είναι γεγονός όμως ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται βάσει ενός στοιχείου που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Το πιο καλό θα ήταν η απλοποίηση, η απλούστευση. Δεν ξέρω πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό, γιατί ασφαλώς και θα ήθελα να προτείνω μια τεράστια απλούστευση, αλλά αυτό Σημαίνει ότι θα έπρεπε ήδη να υπάρχει μια επιτυχία. Γιατί η πραγματική απλούστευση θα υπάρξει τη στιγμή που οι κανόνες θα αντικατασταθούν από την εμπιστοσύνη και από την δυνατότητα να υπάρξει οικονομική και πολιτική τέτοια πολιτική μεταξύ των κρατών μελών. Στο ενδιάμεσο στάδιο θα πρέπει να προσφύγουμε σε άλλα βήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ τον ε, Σταμαν Κάμφρα, την εισηγήτρια, όλους τους συναδέλφους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. Εντοπίσαμε πάρα πολλά σημεία τα οποία προφανώς δεν θα τα θίξει η αυριανή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε πολλά λοιπόν να κάνουμε για θέματα ιδιοκτησίας και ενισχυμένη συνεργασία σε ό,τι αφορά τα μέτρα, τα χάσμα παραγωγής, της εναρμόνισης των διαδικασιών του παραδόξου αυτού να υπάρχει νομισματική ένωση χωρίς ε, σαφή ε, η αρμοδιότητα για την κατανομή αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για την ε, συμμετοχή σας και πέρα στη συνεδρίαση να σας δώσω κάποια στοιχεία. Το σχέδιο έκθεσης θα εξεταστεί στις 26-27 Ιανουαρίου. Προθεσμία τροπολογιών 5 Φεβρουαρίου. Μπορεί αύριο που θα έχουμε την ανακοίνωση να δείξουμε κάποια ευελιξία. Θα δούμε λοιπόν κατά πόσο θα συμφωνήσουν για κάποιες αλλαγές οι συντονιστές. 26-27 Ιανουαρίου λοιπόν προς το παρόν και 5 Φεβρουαρίου η προθεσμία για τις ε, Ευχαριστώ. Επόμενη συνεδρίαση, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στις 9 το πρωί και το απόγευμα.